Bene, colleghi, buongiorno. Ας ε, ξεκινήσουμε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, ε, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Σήμερα λοιπόν η διερμηνία, τη διερμηνία την έχετε σε όλες τις γλώσσες της Επιτροπής μας. Θα ήθελα επίσης ε, να σας ενημερώσω ότι ως συνήθως η Επιτροπή αυτή μεταδίδεται διαδικτυακά. Πάμε λοιπόν στην ανταλλαγή απόψεων με τον Σάιμον Κόβενι, τον Ιρλανδό Υπουργό Γεωργίας, Επισητισμού και Θαλάσσης, Προεδρεύοντα του Συμβουλίου για θέματα γεωργίας και προφανώς η συζήτηση θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Γνωρίζετε ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα αλλά και για το σύνολο της Επιτροπής ε, να έχουμε κοντά μας ε, τον Υπουργό ε, ο οποίος είναι αρμόδιος και είναι και, υπήρξε και συνάδελφός μας ιδιαίτερα ικανός λοιπόν και πρώην συνάδελφος γιατί όπως θα θυμάστε ο Σάιμον ήταν ευρωβουλευτής κατά την προηγούμενη θητεία του Ευρωκοινοβουλίου και το γεγονός αυτό αναμφίβολα επηρεάζει θετικά τις ε, σχέσεις ε, που υπήρξαν ε, με τη δική μας την Επιτροπή, ανάμεσα στην Προεδρία και τη δική μας την Επιτροπή. Η Ιρλανδική Προεδρία λοιπόν υλοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Η Επιτροπή Γεωργίας, αγαπητέ Σάιμον, την προηγούμενη εβδομάδα ενέκρινε τη δική σας τη θέση για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και αυτό σε, όλα τα, σε όλους τους νομοθετικούς φακέλους, τους σημαντικούς. Ε, προφανώς λοιπόν ε, ετοιμαζόμαστε για την Ολομέλεια στα μέσα Μαρτίου. Εκεί θα λάβουμε, ελπίζω με πλειοψηφία, την εντολή διαπραγματεύσεων και έτσι αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι τριμερείς επαφές με την Ιρλανδική Προεδρία. Υπάρχει προφανώς αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που θα είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων για τι δημοσιονομικέ προοπτικέ. Αυτό το θέμα μα απασχολεί πάρα πολύ και στι 7 και 8 Φεβρουαρίου ελπίζουμε οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να συμφωνήσουν επ' αυτού του θέματο. γιατί όσον αφορά τουλάχιστον τι δικέ μα τι διαπραγματεύσει, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε αν δεν γνωρίζουμε ακριβώς τον προϋπολογισμό, το ύψος του προϋπολογισμού για την κοινή γεωργική πολιτική. Και εκ μέρους λοιπόν των συναντέλφων θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Ιρλανδική Προεδρία γιατί κατάρτισε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα, πολύ σημαντικό και εμείς ε, θα εργαστούμε με ζήλο για να επιτύχουμε, αν βέβαια το κατορθώσουμε, μια πολιτική συμφωνία που θα αφορά στους ε, φακέλους της κοινή γεωργικής πολιτικής. Να επιτευχθεί συμφωνία κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής ε, Προεδρίας. Αυτά όσον αφορά τις ε, άμεσες ενισχύσεις. Το πρώτο, τον πρώτο από τους τέσσερις νομοθετικούς φακέλους. Επίσης, την ε, Δευτέρα και την Τρίτη, όπως ξέρετε, τοποθετηθήκαμε σε σχέση με τις εργασίες της Επιτροπής Γεωργίας για τις ε, τροπολογίες, τις τροποποίησεις ε, της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αγαπητέ Σάιμον, σου δίνω τώρα ευθύ αμέσω το λόγο και αρχίζουμε επίση να καταγράφουμε του ενδιαφερόμενου να λάβουν ε, το λόγο. Προφανώ προηγούνται οι συντονιστέ ε, των ε, πολιτικών ομάδων και μετά η συζήτηση είναι ανοιχτή. Σάιμον, έχει το λόγο. Καλή αρχή, βλέπω να χαμογελάνε οι βουλευτές. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Πάολο, πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω για την υποδοχή που μου επιφυλάξατε. Βλέπω πολλούς παλιούς συναδέλφους εδώ. Έχω περάσει πολλές ε, ώρες εδώ στην ε, συνεδριά της ομάδας μας και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Χαίρομαι που μπορώ να είμαι πάλι μαζί σας ως ε, Ιρλανδός Υπουργό Γεωργίας ενώπιον της Επιτροπής Γεωργίας. Φυσικά εκπροσωπώ και το Συμβούλιο λόγω της Ιρλανδικής Προεδρίας. Ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι μαζί σας. Είναι σχεδόν 40 μέρες ακριβώς από τότε που η Ιρλανδία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι για την ευκαιρία να αναφερθώ στα σχέδια της Ιρλανδικής Προεδρίας για την κοινή αγροτική πολιτική και ιδιαίτερα τη μεταρρύθμισή της, αλλά και για άλλα συναφή θέματα. Έχουμε ενώπιόν μας πολύ σημαντικές προκλήσεις στο επόμενο εξάμεινο ή πεντάμινο πια της Ιρλανδικής Προεδρίας που απομένει για να μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μετά από τις ε, συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα για τη μεταρρύθμιση κοινή αγροτική πολιτική. Προτού μπω σε λεπτομέρειε για το θέμα αυτό, να σταθώ λιγάκι στι γενικέ προτεραιότητε τη Ιρλανδική Προεδρία και να αναφερθώ κάπως σε κάποιες ε, νομοθετικές προτάσεις που μάλλον θα εμφανιστούν στους επόμενους μήνες. Η κύρια κατεύθυνση της Ιρλανδικής Προεδρίας μπορεί να συνοψιστεί με τις τρεις λέξεις σταθερότητα, ε, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Μέσα στη στρατηγική της Ευρώπης 2020, για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ανάκαμψη από την χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που αντιμετωπίσαμε, με εστίαση στη βελτίωση της συνολικής και παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πρόθεσης οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτή είναι μια επιταγή η οποία διατρέχει όλες τις ενέργειες της Ιλλανδικής Προεδρίας. Στον τομέα της γεωργίας αυτό σημαίνει ότι οι προτεραιότητές μας θα πρέπει να είναι η θέσπιση συνθήκων για ανανεωμένη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε σχέση με τη μεταρρύθμιση κοινή αγροτική πολιτική. Όπω και για τα άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, η Κομισιόν προτίθεται να παρουσιάσει προτάσεις για το φυτογειονομικό ε, ή φυτογειονομικά θέματα που αφορούν τις καλλιέργειες αλλά και τις ζωικές ε, και τις ε, εκτροφές ζώων. Η Ιρλανδική Προεδρία επίση είναι έτοιμη να ξεκινήσει συζητήσει στο Συμβούλιο για τα θέματα αυτά για να υπάρξει μεγαλύτερη δυνατή πρόοδο μέχρι το τέλο Ιουνίου. Ένα βασικό στοιχείο αυτού του πακέτου είναι η πρόταση για ένα κανονισμό για, τη, για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που θα δημοσιευτεί το Φεβρουάριο. Η Ιρλανδία θέλει να δώσει προτεραιότητα στη συζήτηση αυτή ώστε να μπορέσει μέχρι το τέλος του 2013 να εγκριθεί αυτό το νομοθέτημα. Σίγουρα έχουμε μεγάλες διαδικαστικές προκλήσεις σε σχέση με το πακέτο αυτό. Τα στοιχεία των δαπανών για τα θέματα τροφίμων και ζωοτροφών συνδέονται με τις δημοσιονομικές προοπτικές και όλα αυτά θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ από τις αρχές του 2014. Η Ιρλανδική Προεδρία θα συνεργαστεί με το Συμβούλιο για να γίνει αυτό πραγματικότητα και ελπίζω και η Επιτροπή σας επίσης. Η διαπραγματεύση για μια νομικά δεσμευτική ε, πρόταση επίσης επίκυνται για το πρώτο εξάμεινο του 2013. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε για τη δασική πολιτική ε, τις προτάσεις μας σε μια υπουργική διάσκεψη στο Συμβουλίο των Υπουργών. Ο στόχος μας είναι να έχουμε μια απόφαση η οποία θα επιτρέψει την ε, βιώσιμη διαχείριση των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αποτελέσει ένα ορόσημο προς την κατεύθυνση αυτή η Ιλλανδική Προεδρία. Θα συμβάλλει φυσικά σε όλα αυτά και η Κομισιόν θα δημοσιεύσει και μια στρατηγική για τα δάση το επόμενο, στους επόμενους μήνες, ώστε να τεθούν οι βάσει για μια βιώσιμη και αηφόρο διαχείριση των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να συνεχιστούμε να τα διαχειριζόμαστε, ιδίω η ευθυγράμμιση τη νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συνθήκε Λισαβόνα. Η δική σα συνεργασία είναι κεφαλαιώδη για να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτού του φακέλου στου επόμενου μήνε και υπάρχουν κάποια θέματα φυσικά τα οποία μπορεί να μα απασχολήσουν στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Για τη μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική. Στρέφομαι στις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας για τη μεταρρύθμιση αυτή. Ο στόχος μου είναι να περατωθεί η έγκριση της θέσης του Συμβουλίου και, της, ε, και η διαπραγματική αυτή εντολή στο τέλος του Μαρτίου. Αυτό θα οδηγήσει σε διαθεσμικό διάλογο με την ελπίδα να υπάρξει μια συνολική απόφαση στο τέλη Ιουνίου ή δυνατόν. Δεν υποτιμώ τη σημασία του εγχειρήματο που έχουμε ενώπιόν μα. Είναι πάρα πολύ φιλόδοξη η στόχη αυτή. Θα χρειαστεί έντονη προσπάθεια από όλου και διάθεση συμβιβασμού. Έχουμε μια προσέγγιση η οποία δεν μπορεί να προχωρήσει με βραδεία, με βραδέα βήματα μονάχα. Θα πρέπει να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια γενική συνένεση ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με ταχύτερα βήματα και να ξεπεράσουμε την συνηθισμένη διαδικασία του τριγωνικού διαλόγου και μόνο. Τρία πράγματα πρέπει να γίνουν για να υπάρξει συμφωνία. Καταρχήν, συμφωνία για τι πολιετή δημοσιονομικέ προοπτικέ το ταχύτερο δυνατό. <clears throat> Η ελπίδα μου είναι ότι αυτό θα γίνει στην στο τέλο τη επόμενη εβδομάδα, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε σαφεί ενδείξει σε σχέση με το συνολικό ποσό το οποίο θα είναι διαθέσιμο για την κοινή αγροτική πολιτική ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε στου επιμέρου κανονισμού και κανόνε και πολιτικέ για την γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να δαπανηθούν τα χρήματα αυτά με τον πιο αποδοτικό δυνατό τρόπο. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρξει στου επόμενου δύο μήνε ταχεία πρόοδο σε εκρεμή θέματα ακόμα στο Συμβούλιο. Και τρίτον, και τα τρία βασικά θεσμικά όργανα, Κομισιό, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, θα πρέπει ενεργά να αναζητήσουν αποδεκτές συμβαστικές λύσεις για όλα αυτά τα θέματα. Προσωπικά είμαι αισιόδοξο για το πρώτο από αυτά τα τρία θέματα, όπω είπα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό σημείο το ότι ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Φαν Ρομπάι, αποφάσισε και δήλωσε ότι υπάρχουν καλέ προοπτικέ συμφωνίε για τι πολιετή δημοσιονομικέ προοπτικέ, στη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο τέλο τη επόμενη εβδομάδα. Το Συμβούλιο Γεωργία βέβαια και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταγράψουν προσεκτικά τα, τα πορίσματα της διάσκεψης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για το Συμβούλιο, για μένα, η βασική γραμμή είναι ότι πρέπει να έχουμε ταχεία πρόοδο σε όλα τα θέματα που ακόμα εκκρεμούν. <clears throat> Υπάρχουν 30 ή παραπάνω ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα οποία εκ τη φύση του είναι αυτά που ήταν τα πιο δύσκολα για διαπραγματεύσει μέχρι στιγμή. Παραμένουν πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν και είμαι πλήρω δεσμευμένο στο να μπορέσουμε να περατώσουμε τη διαδικασία αυτή και να καθορίσουμε τη θέση μα στο ταχύτερο δυνατό. Ελπίζω ότι το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο το Συμβούλιο θα έχει μια σαφή θέση για όλα αυτά τα θέματα. Θα εκφραστεί αυτή η θέση στο Συμβούλιο το εαρινό του Μαρτίου και θα είναι σαφή η θέση μα μέχρι το τέλο Μαρτίου. Αυτό παραλληλίζεται σε μεγάλο βαθμό, είναι παράλληλο χρονικά με το χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κινείται προς την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Οι συναδέλφοι μου στο, Υπουργείο, <clears throat> στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας είναι σαφώς δεσμευμένοι να υπάρξει μια θετική συζήτηση στο Συμβούλιο ήδη αυτή τη βδομάδα. Και επίσης υπάρχει θέληση συμβιβασμού από όλους τους εμπλεκόμενους στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας. Πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε και αυτή η θέληση για συμβιβασμούς οφείλεται και στην θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον ε, τρόπο με τον οποίο υπεστήριξε ένθερμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λύσεις για την μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής και την μεγάλη προσπάθεια που έχουν κάνει οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αναγάγουν 8.000 και πάνω τροπολογίες σε ένα πιο ε, λογικό αριθμό προτάσεων και κειμένων που μπορούν να αντανακλούν τη θέση του Κοινοβουλίου. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα τελείωσε αυτή η διαδικασία από την Επιτροπή σα Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Ντεκάστο, τον πρόεδρό σας, τους συζητητέ, συντονιστές και σκιώδεις όλους τους συναδέλφους ουσιαστικά για το τεράστιο αυτό έργο που έχει επιτευχθεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς το Συμβούλιο και το τόνισα και εγώ προς τους συναδέλφους μου. Ελπίζω το Συμβούλιο τώρα θα κάνει κάτι αντίστοιχο με την τεράστια προσπάθεια του Κοινοβουλίου για να μπορέσει να πέρατωθεί αυτή η διαδικασία μέχρι το τέλος Μαρτίου. Εγώ κατέγραψα τις απόψεις του Κοινοβουλίου μέσα από τις τροπολογίες που έχουν διατυπωθεί. Ενθαρρύνομαι από το γεγονός ότι σε πολλούς τομείς υπάρχει σύμπνοια, υπάρχει μια κοινή προσέγγιση μεταξύ των δύο θεσμικών αυτών οργάνων. Παραμένουν φυσικά χώροι και περιοχές όπου αποκλίνουν οι απόψεις των διοθεσμικών οργάνων. Εγώ προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε περισσότερο τις απόψεις μας. Ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι οι διερευνητικές συνομιλίες που θα αρχίσουν ε, συντόμως και φυσικά και μαζί με την Κομισιόν για να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε ορισμένες τεχνικού χαρακτήρα τροπολογίες και να προετοιμαστούμε για τον τριγωνικό διάλογο. Έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι αυτή η διαδικασία θα επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις από τη στιγμή που υπάρχει και η εντολή στο Συμβούλιο για να ξεκινήσει αυτή η διαπραγμάτευση. Εάν συμφωνήσετε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο μέχρι το τέλος Ιουνίου, αυτό προϋποθέτει ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια ιδιαίτερα εύκαμπτη διαδικασία τριγωνικού διαλόγου και στις άτυπες επαφές που ε, συνδέονται με τον τριγωνικό διάλογο. Ελπίζω ότι η Επιτροπή σας θα δεχτεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ξέρω ότι ο πρόεδρος σας είναι διαθέσιμος να ακολουθήσει μια τέτοια διαδικασία για έγκαιρη απόφαση και εγώ θα συνεργαστώ μαζί του για τα θέματα αυτά. Εν κατακλείδη. Τόνισα ότι οι προτάσεις μας ε, καθοδηγούνται από τους στόχους της Ευρώπης 2020. Μια ευφυής, περιεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό είναι και μια σαφή πρόκληση για την κοινή αγροτική πολιτική. Πιστεύω ότι μπορούμε να αδράξουμε αυτή την πρόκληση και αυτό για δύο λόγου. Πρώτα απ' όλα, γιατί οι γενικοί στόχοι που αναφέρθηκαν από την Κομισιόν στι προτάσει, μια βιώσιμη παραγωγή τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βιώσιμη διατήρηση των φυσικών πόρων και εξισορροπημένη ανάπτυξη στον αγροτικό κόσμο, όλα αυτά συναρμόζονται απόλυτα με τους στόχου της Ευρώπης 2020. Είναι στόχοι που όλοι μας και στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζουμε πλήρως. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η κοινή αγροτική πολιτική έχει ένα πολύ θετικό ιστορικό. Έχει υποστηρίξει τον εξυγχρονισμό του ευρωπαϊκού αγροτικού τομέα έχει εξασφαλίσει ότι ο τομέα αυτό μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την βιώσιμη και ε, ποιότητα παραγωγή τροφίμων. Ελπίζουμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική θα εξακολουθήσει να κάνει αυτή τη σύμβολη και στο ε, διάστημα μέχρι το 2020 και επέκεινα. Γι' αυτό θα ήθελα όλοι να το έχουμε αυτό στο μυαλό μα, αντιμετωπίζοντα την πρόκληση μια συμφωνία για τη μεταρρύθμιση κοινή αγροτική πολιτική. Ότι είναι στο συμφέρον όλων των Ευρωπαίων και όχι μονάχα Προ προς το συμφέρον της αγροτικής κοινότητας να υπάρξει μια συμφωνία για τα θέματα αυτά. Ελπίζω ότι όλα αυτά θα δείξουν το πόσο κατεπίγουσα είναι η ανάγκη να έχουμε μια συμφωνία και θα οδηγήσει και σε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα για συμβασικέ λύσει και αποφασιστικότητα να πετύχουμε στο εγχείρημα αυτό. Είμαι έτοιμο να καθοδηγήσω αυτή τη διαδικασία στο Συμβούλιο και να συνεργαστώ με τον κύριο Δεκάστρο, με του συγητέ τους συντονιστές και τα μέλη της ε, Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή τη διαδικασία και από άλλες επιτροπές. Μαζί μπορούμε όλοι να θέσουμε τα θεμέλια για τις μελλοντικέ αυτές εξελίξεις για τον αγροτικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον τρόπο αυτό, κατά την άποψή μου, θα καταδείξουμε ότι οι θεσμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν τίθεται σε δοκιμασία, μπορούν πράγματι να δώσουν καρπού και να επιτύχουν στα εγχειρήματα αυτά. Πριν από τι ερωτήσει και τα σχόλια, θα ήθελα να κάνω μια τελευταία παρατήρηση. Δεν έχουμε ξανακάνει ποτέ κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Δεν υπήρξε ποτέ μια τόσο πολύπλοκη συζήτηση και διαδικασία συναπόφασης στα πλαίσια τόσο πολυπλόκων θεμάτων μέσα στο στενό χρονικό διάστημα που έχουμε τώρα ενώπιόν μας. Αλλά ο χρόνος είναι στο, στην πλευρά μα, διότι υπάρχει αυτό το παράθυρο ευκαιρία για το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να μπορέσουν να περατώσουν αυτή τη διαδικασία. Σχεδόν τέσσερα χρόνια έχουμε δαπανίσει συζητώντα για τη μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική. Υπήρξαν πολιτικέ συζητήσει μεταξύ βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Υπουργών για τα τελευταία δύο χρόνια. Αν δεν επιτύχει το εγχείρημα αυτό μέσα στου επόμενου πέντε ή έξι μήνε, είναι πολύ ρεαλιστική η πραγματικότητα και η προοπτική ότι μπορεί μέσα στην τρέχουσα θητεία αυτού του κοινοβουλίου να μην ευδοκιμήσει αυτό το εγχείρημα, γιατί του χρόνου όλοι θα είσαστε στις υποψήφιες στις εκλογές. Το Σεπτέμβριο ήδη του 2013 θα γίνουν εκλογέ στη Γερμανία που έχουν μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό τονίζω ότι υπάρχει τώρα μια ευκαιρία να κλείσουμε αυτά τα θέματα. Έχουμε μια Επιτροπή Γεωργίας και ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θέλει πράγματι να επιτευχθεί μια λύση για όλα αυτά τα θέματα της μεταρρύθμισης στα αγροτικά θέματα και έχουμε και ένα συμβούλιο που θέλει ακριβώς το ίδιο. Και έχουμε και μια προεδρία που είναι φιλόδοξη, θέλει να προωθεί στα θέματα αυτά για να υπάρξει μια λύση η οποία θα είναι έγκαιρη αλλά όχι βεβαιασμένη και αποτελεσματική. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, κατά την άποψή μου, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν έχουν δείξει την απόδοση που θα θέλαμε όλοι μας για πάρα πολλούς τομείς. Και αυτό είναι μια ευκαιρία να καταδείξουν ότι μπορούν να διεκπαιρεώσουν ένα σημαντικό θέμα και να δείξουν ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει κάποια ελπίδα και κάποια σταθερότητα στον αγροτοτροφημικό τομέα τα επόμενα χρόνια. Μαζί σας νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό πραγματικότητα και αναμένω τώρα τα ερωτήματά σας και τα σχόλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάιμον. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να αρθούμε στο ύψος ε, των περιστάσεων, των ευθυνών μας. Και νομίζω αυτό σαφώς και μπορούμε να το πράξουμε και θέλουμε να το πράξουμε. Για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο έχουμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικές προκλήσεις και είμαι σίγουρος ότι θα εργαστούμε εντατικά με το Συμβούλιο για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό το φιλόδοξο στόχο μας. Και με τον τρόπο αυτό θα εξαλειφθούν και όλες οι ερμηνείες ε, που δόθηκαν για τις ε, εργασίες μας ε, από κάποιο μέσο ενημέρωση, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα τρυφερό, θα μου επιτρέψετε να πω, με το Κοινοβούλιο. Από ε, τα Λεχτέντα διαβλέψαμε την θέλησή σας, απαρασάλευτη θέληση, να συνεργαστείτε μαζί μας. Και έτσι λοιπόν θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους συντονιστές των ομάδων. Ξεκινώ με το ΕΛ και τον κύριο Άλμπερτ Έσ. Αλμπέρτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζουμε κύριε Υπουργέ. Αγαπητέ Σάιμον, χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθες κοντά μας και εγώ προσωπικά χαίρομαι πολύ που η Ιρλανδική Προεδρία αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή έχει αναλάβει την ευθύνη να διαμορφώσει τη μελλοντική γεωργική πολιτική στην Ευρώπη. Βεβαίως ε, όλοι μας με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από το Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας. Γιατί χωρίς ε, χρηματοδότηση δεν μπορούμε να αποφασίσουμε καταληκτικά. Ελπίζω λοιπόν την άλλη εβδομάδα να καταστεί δυνατόν να υπάρξει ένα συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πλαίσιο για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, που επισήμανες ότι εμείς ως Κοινοβούλιο εργαστήκαμε αποτελεσματικά και μέσα στα χρονικά πλαίσια που είχαν προβλεφθεί για μας και διορτώμε κατά πόσο είναι δυνατόν μια διαδικασία με πάνω από 7.000 τροπολογίες να ε, προχωρήσει μια τέτοιου είδου διαδικασία. Απευθύνομαι εδώ στη διοίκηση και της αποδίδω τα εύσημα γιατί πραγματικά κατόρθωσε ε, την προηγούμενη εβδομάδα να ψηφίσουμε και δεν είναι αυτονόητο αυτό, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσον αφορά το προσωπικό ε, δεν είμαστε, δεν μιλάμε επίση ώρες. Η Κομισιόν έχει πάρα πολλούς συνεργάτες και το Συμβούλιο στα κρατημέλη. Εμείς περιορισμένο αριθμό συνεργατών και παρόλα αυτά τα καταφέραμε μια χαρά. Ελπίζω λοιπόν ότι εφόσον είναι γνωστή η θέση του Κοινοβουλίου Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε από κοινού το Συμβούλιο να ε, σχεδιάσουμε αποτελεσματική πολιτική για το χρονικό διάστημα μετά το 2014. Και θέλω τη γνώμη σου. Η Ιρλανδική Προεδρία το αργότερο τον Ιούνιο θα ολοκληρώσει τις εργασίες της ε, και νομίζω το πολύ πολύ που μπορεί να πετύχει είναι ένα πρόγραμμα εργασίας για μέχρι το τέλος ε, του 2014. Καθαρά ρεαλιστικά τη νέα αγροτική πολιτική θα μπορούμε να εφαρμόσουμε την πρώτη πρώτη του 2015. Το 2014 θα το χρειαστούμε έτσι ώστε η νέα αγροτική πολιτική να εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη. Ε, προσυπογράφω όλα αυτά που είπες. Ε, πράγματι όλους εμάς μας ενδιαφέρει μια ανταγωνιστική βιώσιμη γεωργία στην Ευρώπη και πρέπει αυτό να το επαναλαμβάνουμε στην κοινή γνώμη Οποτεδήποτε γίνεται η συζήτηση γιατί η γεωργική πολιτική καταλαμβάνει ένα τόσο μεγάλο κομμάτι των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να λέμε αυτό οφείλεται ότι η πολιτική, η κοινωνική, η ερευνητική, η αμυντική πολιτική, αυτές όλες δεν είναι τόσο εξευρωπαϊσμένες όσο η γεωργική πολιτική. Αν ήταν στο ίδιο βαθμό ευρωπαϊκές θα συνέβαινε ίσως και για αυτές το ίδιο. Άρα δηλαδή οφείλουμε να υπογραμμίζουμε ότι τα κονδύλια που χρησιμοποιούνται για την γεωρική πολιτική ωφελούν 500 εκατομμύρια καταναλωτές. Εγώ είμαι αισιόδοξο ότι υπό την Ιρλανδική Προεδρία θα προχωρήσουμε ικανοποιητικά και ε, σου εύχομαι καλή τύχη. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ, ε, Άλμπερτ, ο κύριος ε, Κάπουλα Σάντος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να χαιρετήσω τον Υπουργό Σάιμον Κόβενε, Καλώς ήρθατε και καλή επιτυχία για την Προεδρία. Είμαι συντονιστής των σοσιαλιστών και εισηγητής για τη σχετική έκθεση και δηλώνω ικανοποιημένος που είναι η σειρά της Ιρλανδικής Προεδρίας. Δεν υπάρχει καλύτερη χώρα γιατί έχει ιδιαίτερη για τα γεωργικά ζητήματα και θα καλύψει καλύτερα τις προσδοκίες μας σε αυτό το τομέα. Συμφωνώ με τις προτεραιότητες που θέσατε και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι δείχνατε αποφασισμένοι και εμείς εξίσου αποφασισμένοι είμαστε, σας διαβεβαιώ. Έχουμε αναλάβει σοβαρότατη δέσμευση για να καταλήξουμε συμφωνία επί Ιρλανδικής Προεδρίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέδειξε ένα συμβαστικό πνεύμα στις διαβουλεύσεις που έκανε και ευελπιστώ να επικρατήσει το ίδιο συνενετικό πνεύμα και στο Συμβούλιο τους επόμενους μήνες. Σε σχέση με τις δύο εκθέσεις όπου είμαι εισηγητής, καταφέραμε να ε, καταλήξουμε τελικά σε 75 τροπολογίες από τις 3.000 που είχαμε αρχικά. Ε, με ιδιαίτερη προσοχή εξετάστηκαν και από τους σκιώδεις εισηγητές και στη ψηφοφορία τηρήθηκαν τα συμπεφωνημένα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τους σκιώδεις εισηγητές και ως επιτοπλίστων εγκρίθηκαν ε, με συντριπτική πλειοψηφία αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες. Το Συμβούλιο γνωρίζει πολύ καλά τις θέσεις μας και θα ήθελα, Υπουργέ, για να μην ε, μακρηγορώ, γνωρίζοντας λοιπόν τις θέσεις του Κοινοβουλίου, θα ήθελα να μας πείτε σε ποια ζητήματα θεωρείτε εσείς ότι θα ανακύψουν σοβαρότερες ε, δυσκολίες με τρόπο ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε επιμακρών αυτά τα ζητήματα, και να προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση. Εγώ προσωπικά, θα πω κλείνοντα, ε, είμαι στη διάθεσή σας για να κάνουμε όποιε άτυπε επαφέ, κρίνετε εσείς απαραίτητες. Νομίζω ότι πέρα από τις επίσημε διαπραγματεύσεις, ο καιρός επιτάσσει μεγαλύτερη ευελιξία και διαλλακτικότητα για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα ε, χαίρομαι επίσης που αναγνωρίσατε την αποτελεσματικότητα των εργασιών του Κοινοβουλίου και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι του επόμενους μήνες. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Λουίς. Ε, η Μπρίτα ε, από τους Φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εγώ χαίρομαι που μπορώ να σας υποδεχτώ εδώ. Να, εδώ είμαι από την πλευρά της ομάδας των φιλελευθέρων. Ξέρουμε όλοι πόσο μεγάλο είναι αυτό το εγχείρημα που έχουμε ενώπιόν μας και πόσο σύντομος είναι ο χρόνος στον οποίο πρέπει να επεξεργαστούμε όλα αυτά τα θέματα. Εμείς εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Ιρλανδική Προεδρία είναι έτοιμη να ανοίξει νέους δρόμους για τα θέματα αυτά και εμείς είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε το ταχύτερο σε μια συμφωνία. Όπως είπατε, ο χρόνος μας πιέζει Ξέρουμε ότι ο Ιρλανδικός λαός είναι γνωστός για την ανθεκτικότητα και την επιμονή του και ξέρουμε ότι αυτό θα σημαίνει ότι εσείς μπορείτε να πείσετε το Συμβούλιο αυτά τα 30 εκκρεμή θέματα να τα κλείσει επιτέλους, να καταλήξει σε μια συμφωνία. Και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά έχουμε μια πολυπληθώρα απόψεων μεταξύ μας, αλλά μπορούμε όλοι να είμαστε ικανοποιημένοι με την λύση στην οποία καταλήξαμε μετά από πολλές διαπραγματεύσεις. Ελπίζω ότι το ίδιο πράγμα θα μπορέσει να γίνει και στο Συμβούλιο, ώστε να μπορέσει να προέλθει μια λογική εντολή διαπραγμάτευσης για το τριγωνικό διάλογο. Εμεί ω Κοινοβούλιο θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να μπορέσει αυτός ο τριγωνικό διάλογο να ευδοκιμήσει και να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λύση η οποία θα είναι ικανοποιητική για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και εκ μέρους των ε, Πρασίνων ο Μάρτιν. Κύριε Υπουργέ, και εγώ θα ήθελα να σας χαιρετήσω θερμά εκ μέρους των ε, Πρασίνων. Νομίζω συμφωνούμε όλοι μας. Ε, έχετε καταρτήσει ένα ιδιαίτερο φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα που είναι απαιτητικό και για μας. Δεν δεσμευτήκαμε ακόμα, αλλά σύντομα πρέπει να το κάνουμε. Βεβαίως Ίσως μπορείτε να επιδείξετε κάποια ευελιξία ε, και όχι να ε, οργανώσετε τις ε, συναντήσεις στο πλαίσιο ενός ε, άκαμπτου τριλόγου. Θα μας το πείτε την επόμενη εβδομάδα. Πάρα πολλά εξαρτώνται από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι θα πράξουν αποφάσεις που θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις. Ως προς τις περικοπές, στον πρώτο και στο δεύτερο πυλώνα υπάρχει μια ανισορροπία στις περικοπές και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Εντάξει, ε, υπάρχουν περικοπές και στον πρώτο πλάνο, όχι τόσο μεγάλες όσο στο δεύτερο. Στο δεύτερο κυρίως ε, σημαντικές περικοπές και αυτό φύγει πολλά κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να μεριμνήσετε έτσι ώστε να μην παραμείνει αυτή η ανισορροπία. Ο κύριος Βαν Χομπέι έχει εντάξει πολλά στους ε, συμβιβασμούς που κατ' όμως δεν είναι δικές του αρμοδιότητες. Είναι αρμοδιότητες στον τομέα της ε, γεωργίας. Με εντυπωσιάζει λοιπόν που ο κ. Βαν Ρομπέη ανέλαβε θέματα που κατ' ουσία είναι θέματα ε, του ε, Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και όλα αυτά δεν διευκολύνουν τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά και ανοιχτά θέματα. Εμείς θα πούμε τη θέση μας, θα φανεί η θέση μας όταν θα έχουμε ψηφίσει. Ε, στις ε, διαπραγματεύσεις ε, σημαντικό ρόλο έπαιξε οι ιστορικές αυτές πληρωμές τις οποίες απεχαιρετήσαμε διαπαντός η Γερμανία εισήγαγε ένα περιφερειακό μοντέλο και αυτό αποτελεί τη βάση έτσι ώστε σε τελική ανάλυση το σύνολο των κρατών της Ευρώπης να αποκτήσουν την ίδια ανταγωνιστικότητα και ισότητα ευκαιριών. Νομίζω λοιπόν πρέπει όλοι μας να είμαστε λίγο περισσότερο φιλόδοξοι. Αυτό αφορά την προσαρμογή των πληρωμών στην Ευρώπη. Πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα γιατί αλλιώς ε, θα χάσουμε την υποστήριξη ε, των ε, υποψήφιων κρατών. Και αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι δεν πρόκειται μόνο για την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας. Η κοινή γνώμη απαιτεί στις μεταρρυθμίσεις να θίξουμε και το θέμα της προστασίας, της κλιματικής προστασίας ε, και αυτά όχι μόνο κάτω από επικεφαλίδες, γιατί εντωμεταξύ όλοι είναι για το πρασίνισμα. Όμως, αν δει κανείς λιγάκι τι σημαίνει πρασίνισμα, αυτό ε, είτε αφήνεται στη διακριτική ευχαίρεια του καθενός ή ε, μεταβιβάζεται στα κράτη-μέλη. Εμείς αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Πρέπει να εξηγήσουμε στην κοινή γνώμη ότι τα χρήματα που δίδονται για το πρασίνισμα κατ' ουσίαν αποτελούν επιβράβευση για την ενασχόληση με το περιβάλλον. Εμείς ως πράσινοι επιθυμούμε να ε, κινητοποιήσουμε καταστάσεις ε, στον τομέα του περιβάλλοντος. Ε, κάποιες τροπολογίες μας δεν μπορούσαμε να τις περάσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω η κοινή γνώμη περιμένει να κάνουμε βήματα προς μια βιώσιμη γεωργία η οποία τελικά θα εφαρμοστεί από τα κοινοτικά όργανα. Jim Nicholson, επόμενος ομιλητής, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα με τη σειρά μου να καλωσορίσω τον Προεδρεύοντα του Συμβούλιο, τον Υπουργό Κόβενε. Καλή επιτυχία για τις επόμενους πέντε μήνες, διότι πέρασε ο πρώτος είδε και θα είναι πολύ εντατική η ρύθμη, φαντάζομαι, προς το τέλος, όπως πάντα, αλλά νομίζω ότι θα είμαστε όλοι σε θέση να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Στην, ε, α, στα εναρκτήρια σχόλιά σας μιλήσατε για πολύ σημαντικούς ε, συμβιβασμούς. Ε, ξέρετε, είναι η ειδικότητά μας εδώ οι συμβιβασμοί και προσπαθούμε <coughs> να βρούμε συμβαστικές λύσεις σε τομείς όπου αποκλίνουν σημαντικά οι απόψεις μας. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι θα ανταποκριθεί και το Συμβούλιο, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, διότι ε, σε όλες τις επαφές που είχα μαζί τους μου δόθηκε η εντύπωση ότι έχουν ελιπέστατες γνώσεις σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα πολύ δύσκολο έργο για εσά να περάσετε αυτό το μήνυμα, ότι δεν μπορούν να μας πατάνε και να κάνουν ό,τι θέλουν ε, ή ότι είμαστε εδώ για να ακούμε τι έχουν να μας πούν εκείνοι. Όχι, είμαστε ένα σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τη μεταρρύθμιση κοινή γεωργικής πολιτικής. Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω για την επιστημιστική ασφάλεια. Αυτό ήταν το μεγάλο ζητούμενο πριν από δύο-τρία χρόνια. Όλοι γι' αυτό μιλούσαν, όλοι θεωρούσαν ότι είναι καταπληκτική ιδέα. Μπορείτε να μου πείτε πού ακριβώς, πώς με αυτές τις προτάσεις θα κατοχυρώσουμε την επιστημιστική ασφάλεια για το μέλλον, διότι εγώ δεν έχω καταφέρει να βρω κάποιο τέτοιο στοιχείο. Κάθε γεωργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερα παραστατικά και οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, οφείλω να ομολογήσω ότι θα επισύρουν τουλάχιστον ε, ένα επιπρόσθετο 15% και σε κόστο και σε γραφειοκρατία. Οπότε δε... βλέπουμε ότι με τις προτάσεις που εγκρίθηκαν την περασμένη εβδομάδα δεν βελτιώνεται η κατάσταση. Δεν θα είναι μικρότερο το επιπρόσθετο κόστος, ούτε και η επιπρόσθετη γραφειοκρατική διαδικασία. Μας είπαν στην αρχή ότι έπρεπε να δεχθούμε το πρασίνισμα και τον πρώτο πυλώνα για να εξασφαλίσουμε τα κονδύλια. Τώρα τα έχουμε και το πρασίνισμα και το πυλώνα είναι περικόπτουν όμως τον προϋπολογισμό. Με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα, διότι είναι και το κέριο σημείο σε διαπραγματεύσει. Τι θα γίνει με το πρασίνισμα, θα μείνει στον πρώτο πυλώνα, αν περικοπεί ο προπολογισμό ή πρέπει να πάει όπω πιστεύαμε πολλοί από εμά στον πυλώνα 2. Αυτοί οι τομης ε, θα μας απασχολήσουν και θα μας δυσκολέψουν και εσάς και εμάς. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να λειτουργεί επί τόπου η γεωργική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το μεγαλύτερο σφάλμα μας είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε νέα λύση από το βορρά προς τον νότο και από την Ανατολή μέχρι τη Δύση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν λειτουργεί η ίδια λύση για όλους. Θα πρέπει λοιπόν να επιτύχουμε μεγαλύτερη ε, ευελιξία, ούτως ώστε όντως να λειτουργήσει στην πράξη η λύση στην οποία θα καταλήξουμε. Είπατε ότι έχουμε τώρα την ευκαιρία να, κάνουμε, να οικοδομήσουμε ένα σύστημα που θα λειτουργεί. Σας διαβεβαιώ ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να έχουμε τελικά συμφωνία Πρωτού λήξει η Ιρλανδική Προεδρία. Αλλά σας λέω ότι δεν πρόκειται να δεχθώ ούτε ολόκληρη συμφωνία, ούτε τμηματικά μια συμφωνία η οποία δεν θα λειτουργήσει επί τόπου. Εγώ θέλω να αφιερώσω το χρόνο οικονομία να καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία θα λειτουργεί αισίως και για αυτούς που την διαχειρίζονται την νέα πολιτική σε κυβερνητικό επίπεδο, σε, για αυτούς ε, που στην, ε, μέσα στην αγροβιομηχανία θα κληθούν να εφαρμόσουν τη νέα μας πολιτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Τζιμ. Τώρα λοιπόν, ε, εξ ονόματος του αφεντή, συνάδελφος Έλμερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Εγώ αντικαθιστώ τον συνάδελφό μου τον κύριο Άγνιου. Μπορεί να σας ανακουφίζει η απουσία του, αλλά θα προσπαθήσω να καλύψω το κενό. Έχετε μόνο 6 μήνες κύριε Κόβενη για να βελτιώσετε αυτή την εμβαλωματική κατά κάποιο τρόπο πρόταση για την κοινή αγροτική πολιτική. Πού είναι η απλοποίηση, αυτή ήταν ένα στόχο, αλλά την έχουμε χάσει αυτή την έννοια τη απλοποίηση. Πού είναι η μείωση τη γραφειοκρατίας. Είναι πολύπλοκοι κανόνες για τους τομείς οικολογικής εστίασης, διαφοροποίηση, διαχείρισης γεών, διπλή ε, δυνατότητα χρηματοδότησης από τους φορολογούμενους. Πώς κάνει τα πράγματα αυτό πιο απλά ή πιο διάφανα. Δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση καθόλου. Είναι τα ίδια που είχαμε και στο παρελθόν. Το χειρότερο είναι ο προστατευτικός Χαρακτήρα τη ε, πρόταση του κυρίου Νταντέν που θέλει να υποστηρίξει παραδοσιακέ αγορέ όπω αυτή τη ζάχαρης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πληρώνουν, καταναλωτέ πληρώνουν δύο φορέ περισσότερο τη ζάχαρη που θα μπορούσαν να παίρνουν φτηνότερα από όλο. Αυτό οδηγεί σε απώλεια να απασχόλησης στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού. Ο κύριο Σάγνη μου ζήτησε να τονίσω όπω και άλλε φορέ το έχει κάνει το θέμα τη εταιρεία State Line στο Ηνωμένο Βασίλειο θυμίζει τα ερωτήματα που κατέθεσε για τη μεταρρύθμιση τη αγορά ζάχαρη το Νοέμβριο του 2012 που δεν έχουν τύχει απάντηση. Μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι τα ζητήματα αυτά θα αντιμετωπιστούν ταχαίω. Η πρόταση ενώπιών μα, οι προτάσει ενώπιών μα δεν κάνουν τίποτα για να λύσουν τα προβλήματα αυτά. Σε μια στιγμή που οι τιμέ των τροφίμων αυξάνονται, οι προτάσει αυτέ δείχνουν προστατευτισμό, κακοδιαχείριση τη αγορά που επιβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο για 10 χρόνια ακόμα. Σα ζητώ κύριε Κάβενη να χρησιμοποιήσετε την Ελλαδική για να φέρετε και κάποια κοινή λογική στι προτάσει αυτέ και να εξασφαλίσετε ότι σε μια στιγμή που αυξάνονται οι τιμέ και προβλέπονται ελλείψεις τροφίμων, οι γεωργοί δεν περιορίζονται από ένα σύστημα το οποίο περιλαμβάνει αυτές τις τρευλές προβλέψεις για πρασίνισμα. Και ότι οι γεωργοί στη χώρα μου και σε άλλες χώρες που έχουν δηληστήρια ζάχαρης δεν θα χάσουν τις δουλειές τους χάρη, λόγω αυτών των μεταρρυθμίσεων. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Τελείωσε λοιπόν ο γύρος ε, που αφορούσε τους ε, συντονιστές ε, και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Σάιμον για να απαντήσει και κατόπιν θα ξεκινήσουμε με τους σκιώδης ηγητές και όλους τους άλλους που ζήτησαν το λόγο. Σάιμον, έχεις το λόγο. Λοιπόν, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις που μου υποβάλλατε και που ήσασταν ανοιχτοί απέναντί μου. Ε, πολύ καλύτερο αυτό από τις φιλοφρονήσεις. Ε, στα σχόλια του Άλμπερτ να πω. Συμφωνώ μαζί σου ότι την επόμενη εβδομάδα πρέπει να υπάρξει συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να προχωρήσουμε από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Ε, πρέπει να περάσουμε στην ε, τελική φάση των θέσεών μας, να ξέρουμε πόσα χρήματα θα δοθούν ε, για την κοινή γεωργική πολιτική στο πλαίσιο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Κάτω από το πρίσμα των Υπουργών πρέπει να λάβουμε ώστε το δυνατόν περισσότερες αποφάσεις ε, όσον αφορά στην εφαρμογή, στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και όλα αυτά βέβαια σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο λόγω της διαδικασίας συναπόφασης. Όμως την επόμενη εβδομάδα... Ε, θα ληφθούν κάποιες ε, αποφάσεις ε, αυτά θα τα χειριστεί ο κύριος Βαρομπέη. Θα πρόκειται για το πρασίνισμα, για την εξωτερική σύγκληση ανάμεσα σε διάφορες χώρες και τα υπόλοιπα του box αυτού των διαπραγματεύσεων που είμαι σίγουρη ότι όσοι έχετε παρακολουθήσει τη συζήτηση τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μετά λοιπόν από αυτή τη συνάντηση θα έρθει κάποιος από την Κομισιόν που θα μιλήσει για μεταβατικές διατάξεις νομίζω μετά το 2014 νομίζω όλοι δέχονται ότι θα πρέπει να παρεμβάλλετε μία χρονιά, όχι παραπάνω, από τη φάση όπου ε, ολοκληρώνεται η συμφωνία και τη στιγμή που οι χώρες πλέον εφαρμόζουν αυτή την πολιτική. Ε, πολλοί από εσά, ε, ο Τζίμο Ρότζερς και άλλοι, το έθιξαν το θέμα και πράγματι ό,τι και αν κάνουμε εδώ για να αλλάξουμε μια πολιτική καταρχήν πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα κράτη-μέλη έχουν χρόνο να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική. Οι οργανισμοί πληρωμών και όλα τα άλλα πρέπει να λειτουργούν έτσι ώστε η πολιτική να λειτουργεί απλά, να την κατανοούν οι αγρότες ε, και να είναι όλα εφικτά. Δεν μπορούμε να τα βιάσουμε και γι' αυτό λοιπόν και η Κομισιόν δέχτηκε ότι ακόμα ακόμα και αν επιτευχθεί η πολιτική συμφωνία τον Ιούνιο, οι υπόλοιποι έξι μήνε είναι απαραίτητοι για να τεθεί σε ισχύ ένας κανονισμός. Να υπάρχει μια μεταβατική ρύθμιση για το 2014 υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συμφωνία για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και εφαρμογή από το 2015. Νομίζω αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα επί του οποίου εργαζόμεθα αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τώρα στα σχόλια της Λουίζας, ε, κοιτάξτε, ε, χαίρομαι ε, που ε, έχετε αποκομίσει αυτήν την εντύπωση. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά το ρόλο του Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία, όπως επίσης και τα σχόλια που έκανε ο Τζιμ. Ήμουνα τρία χρόνια Ευρωβουλευτής και γνωρίζω πολύ καλά την απογοήτευση που επικρατεί εδώ όσον αφορά την διαδικασία της συναπόφασης. Και αυτό το που έχουμε είναι πράγματι η μεγαλύτερη ευκαιρία ε, συναπόφασης που έχει προσφερθεί όχι μόνο στην Επιτροπή αλλά στο σύνολο του Κοινοβουλίου και ελπίζουμε να στεφτεί τελικά από επιτυχία. Οι τομείς ε, που είναι δύσκολοι, κοιτάξτε, είναι δύσκολο για μένα να σας αναφέρω μια συγκεκριμένη απάντηση από αυτού, διότι το Κοινοβούλιο δεν έχει ολοκληρώσει την διαπραγματευτική του θέση. Νομίζω όμως ότι κάποιοι τομείς που είναι δύσκολο για σας να συμβαστείτε, είναι δύσκολο και για μένα να επιτευχθεί συμφωνία στο Συμβούλιο. Δεν θέλω να υποτιμήσω την πρόκληση για την Προεδρία στο να υπάρξει μια τελική δική της θέση. Υπάρχει διάσταση απόψεων για πάρα πολλά θέματα. Νομίζω όμως, εάν υπάρχει συμφωνία για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα εργαστούμε πολύ σκληρά και υπάρχει υπάρχει ουσιαστική βούληση να καταλήξουμε σε συμβασμό. Βεβαίω με το Κοινοβούλιο θα διαπραγματευτούμε για το πρασίνισμα, την εσωτερική σύγκληση, την υποστήριξη των ε, νέων γεωργών, το περίφημο κάπινγκ ε, ε, και επίσης τη διαχείριση των αγορών, την κοινή οργάνωση αγοράς Υπάρχει διάσταση υπόψεων και στο Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο. Υπάρχουν χώρε που επιθυμούν μια πολύ πιο ελεύθερη προσέγγιση αγορά και άλλε χώρες που ε, ενοχλούνται, αυτές επιθυμούν να ελέγχουν περισσότερο και τι αγορέ ε, και τι ε, τιμέ. Πάντα θα υπάρχει αυτή η προστριβή και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο και φαντάζομαι ότι θα εξακολουθήσει να υπάρχει αυτή η διάσταση απόψεων και όταν αρχίσουν οι διαπραγματεύσει με τα όργανα. Εναπόκειται λοιπόν σε όλου μα να βρούμε μια ε, ρεαλιστική τροχιά. Για τα επόμενα σχόλια, ε, Προφανώ υπάρχει η διάσταση απόψεων και όπω σα είπα αυτή θα επιταθεί. Ο Μάρτιν, Μάρτιν Χάουσλινγκ και πάλι θέλω να πω είναι δύσκολο για μένα να αναφερθώ με λεπτομέρειες στο πρασίνισμα που ξέρω ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα αν δεν υπάρχει ε, διαπραγματική εντολή από το Συμβούλιο. Μπορώ να σας πω τις ε, προσωπικές απόψεις αλλά ξέρετε τι έτσι κάνετε αυτές. Γιατί αυτό που χρειάζεστε είναι μια διαπραγματική, διαπραγματευτική εντολή, ε, απλή, κατανοητή και παράλληλα ε, η συμφωνία σε προτάσεις που έχουν αξία. Ε, να είναι βιώσιμες οι προτάσεις ε, και να έχουν αυτά αποτελέσματα στο θέμα των τροφίμων. Είναι αλήθεια ότι το ελεγκτικό συνέδριο υπολόγισε ότι η εφαρμογή της νέας κάπου όπως την έχει χαράξει η Κομισιόν ίσως οδηγεί σε αύξηση του κόστους κατά 50% και αυτό είναι απαράδεκτο κατά την άποψή μου. Είναι απαράδεκτο και για το Συμβούλιο και είναι απαράδεκτο και για το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν καταθέσατε χίλιες τροπολογίες και γι' αυτό προτείνατε απλούστερη εφαρμογή των προτάσεων από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί από την Κομισιόν. Δεν έχει νόημα να στρέφεστε σε μένα και να ζητάτε την απλούστευση. Για να δούμε λιγάκι ποια είναι η θέση του Κοινοβουλίου για την απλούστευση και έτσι να ξεκινήσετε τις ε, τριμερείς. Εσείς μου λέτε ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι καθοριστική σημασία σε αυτή τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Αν ισχύει αυτό και εσείς έχετε τις ίδιες ευθύνε όπως και εγώ ε, για να υπάρξει απλούστευση και μία ε, λειτουργική πολιτική. Να μιλάμε επίσης όρις και όχι να περιμένετε από μένα τις απαντήσεις και εγώ ε, θα προσπαθήσω να βρω τις καλύτερες απαντήσεις μέσα από διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο να κάνετε κι εσείς το ίδιο και τελικά ελπίζω ότι η δύο αυτές συμβαστικές προτάσεις θα οδηγήσουν σε ένα τελικό συμβασμό που θα ικανοποιεί όλους. Ορισμένες από τις συμβαστικές προτάσεις ε, πράγματι ε, καθοδηγήθηκαν από τους δικούς σας τους συμβασμούς ε, των τελευταίων εβδομάδων. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες από αυτού τώρα, τώρα μα νομίζω είναι σημαντικό να το πει κανείς Ορισμένες λοιπόν συμβαστικές προτάσεις βγάζουν νόημα, άλλες πάλι είναι δύσκολες. Ε, αν ε, δεν υπήρχε η συναπόφαση, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Όσον αφορά τα σχόλια του Τζιμ, είσαι ξεκάθαρος όπως πάντα. Κοίταξε, όσον αφορά την επιστηστική βοήθεια, εγώ προσωπικά ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για το θέμα αυτό. Ε, και επέμεινα στο Συμβούλιο ο Συρλανδός να τεθεί το θέμα. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ουσιαστική γεωργική πολιτική ε, πρέπει να προσφέρει επισητιστική ασφάλεια συμβατή με το περιβάλλον και με την προστασία, κλιματική προστασία. Αλλά να είμαστε ξεκάθαροι. Ε, το 2030 γνωρίζουμε ότι ε, θα χρειάζονται τότε σε παγκόσμιο επίπεδο 40 με 50% περισσότερα τρόφιμα από ό,τι τώρα. Ε, αυξάνεται, υπάρχει δημογραφική ανάπτυξη, περισσότερες ε, εξελίξεις ε, και έτσι λοιπόν η Ευρώπη πρέπει να παίξει και αυτή το δικό της το ρόλο. Είναι πολύ εύκολο να βρει κανείς ε, απαντήσεις ε, για την, σε σχέση με τη βιωσιμότητα. μπορούμε να παράγουμε λιγότερο και να μην ασκούμε πίεση στη γη. Αλλά δεν είναι όμως αυτή η πραγματική πρόκληση. Η πρόκληση είναι πώς θα παράγουμε τρόφιμα με βιώσιμο τρόπο έχοντας κατά νου και όλες αυτές τις ε, προκλήσεις ε, τις πολλαπλούς ε, συμμόρφωσης γιατί το θέμα είναι επειδή υπάρχουν οι προκλήσεις πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές και παράλληλα να παράγουμε περισσότερα τρόφιμα. Περίπλοκη αυτή η πρόκληση και γι' αυτό το πρασίνισμα είναι σημαντικό να είμαστε απλοί να έχει πραγματική αξία το πρασίνισμα, όχι να είναι μια επιφανική διαδικασία. Οι παραγωγοί να θέλουν πράγματι να παράγουν περισσότερο με έναν τρόπο που θα είναι ανταγωνιστικός όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Σημασία έχει πώς μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά και παράλληλα να διαχειριζόμαστε τη βιωσιμότητα ε, με αποδεκτό τρόπο. Αυτή είναι η πρόκληση της ΚΑΠ και αυτό ε, προσπαθούμε να κάνουμε και σε σχέση με τους ε, μηχανισμούς του πυλώνα 2 οι χώρες ε, να έχουν κάποιες προτεραιότητες, οποιασδήποτε και αν είναι αυτές, ε, σε αντίθεση με πιο πολύπλοκους μηχανισμούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πυλώνα 2. Είναι δηλαδή σαν να ζητάμε από τις χώρες στον πυλώνα 2 να δαπάνουν περισσότερα χρήματα, αλλά όταν προσπαθούν να το κάνουν να, τους, να τις εμποδίζουμε στο Συμβούλιο δεν έχουμε βρει ακόμα όλες τις απαντήσεις, αλλά εργαζόμαστε για να τις βρούμε. Και τέλος, όσον αφορά τα σχόλια του Ρότζες, σε, θυμάμαι και εγώ με μεγάλη χαρά από τότε που ήμουν εδώ στο Κοινοβούλιο Ρότζερ. Κοίταξε, εμείς εξτάζουμε τα, θάματα, τα θέματα από τελείω διαφορετικό πρίσμα όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη δική μου άποψη, αξίζει τον κόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει λογική ως προς την παραγωγή τροφίμων, το πώς προστατεύουμε το περιβάλλον, της ε, πόλης μας, γιατί η κοινή γεωργική πολιτική είναι η μόνη οικονομικά κατανοητή πολιτική που έχει λειτουργήσει και εξακολουθεί να αποδίδει. Έχει ελλείψεις, γι' αυτό πρέπει να την βελτιώσουμε. Πρέπει να την απλουστεύσουμε και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ανταγωνιστική τόσο στην αγορά ζάχαρης όσο και σε άλλες αγορές και πρέπει να επωφεληθούμε και από άλλες αγορές που επεκτείνονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πράγματι στο μέλλον πρέπει να προστατεύσουμε τη βιομηχανία ζάχαρης και επίτρεψέ μου να σου πω η Ιρλανδία είναι ειδική για θέματα ζάχαρης. Ε, δεν θέλω τώρα να μπω ε, σε λεπτομέρειες όσον αφορά τις δικές μου προστατικές απόψεις για το καθεστώς της ζάχαρης. Τέτον Λάιλ, κοιτάξτε, δεν έχω λεπτομέρειες να σας αναφέρω, αλλά αν μπορώ να βοηθήσω σίγουρα θα το κάνω. Και δεν θέλω να δώσω υπερβολικές ε, ε, υποσχέσεις. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ε, μπορείτε να επεξεργαστείτε, να το συζητήσετε με την Κομισιόν. Αυτά μπορούσα να πω προς το παρόν και βεβαίως περιμένω να υποβάλλετε και άλλες ερωτήσεις. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε Σάιμον και επίσης σε ευχαριστούμε και για τον τρόπο, τον ξεκάθαρο με τον οποίο αντιμετωπίζεις τις ερωτήσεις. Κύριε Ρούμπιξ, εκ μέρους των ε, κομμουνιστών. Δεν σε είχα δει και σου δίνω μέσα στο λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα συμφωνήσω με κάποιους από τους προαναλύσαντες. που έδειξαν και κάποια κατανόηση σε σχέση με αυτά που είπατε όταν μπήκατε στην αίθουσα. Και εσείς χαμογελούσατε όταν ξεκινήσατε και τα λόγια σας δίνουν την εντύπωση ότι πάρα πολλά πράγματα μπορούν να υλοποιηθούν. Ξέρω ότι δεν εξαρτάται μόνο από εσά και μόνο από το Συμβούλιο, <clears throat> αλλά είμαι πεπισμένος ότι η Ιρλανδική Προεδρία θα χρησιμοποιήσει αυτή την, την κρίσιμη χρονική περίοδο, την τελευταία ευθεία ως το νήμα, για να υπάρξει η σωστή ρύθμιση για την κοινή αγροτική πολιτική. Από ό,τι καταλαβαίνω, η, η Ιρλανδική Προεδρία έχουν δείξει την ικανότητά τους σε δύσκολες χρονικές στιγμές να ακούν τη φωνή των λαών και να δρουν με τέτοιο τρόπο ώστε τα αιτήματα του, του πληθυσμού να γίνονται ακουστά. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε και εμείς ως βουλευτές και ως εκπρόσωποι των λαών να συμβάλλουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και ελπίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσετε και εσείς να δράσετε υποστηρίζοντας τις συμβαστικές λύσεις στις οποίες έχουμε καταλήξει. Εδώ και δύο χρόνια εργαζόμαστε <clears throat> για την κοινή αγροτική πολιτική και έχουν γίνει δεκάδες εκδηλώσεων διαμαρτυρίας είδαμε κόσμο να έρχεται με τα τρακτέρ ενώπιον μπροστά στο κοινοβούλιο, να φωνάζουν, να ρίχνουν γάλα στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, ως εκπρόσωπος της δικής μου πολιτικής ομάδας, της ΓΚΟΕ και ως εκπρόσωπος της Λετωνίας, θα ήθελα να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τις άμεσε πληρωμές, και αυτό αναφέρθηκε και από ορισμένου συναδέλφου προηγουμένω, η τωρινή κατάσταση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι αποδεκτή. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση <clears throat> θα πρέπει να έχει το χαρακτήρα της δικαιοσύνης. Μου με ρωτάνε πάντα οι ψηφοφόροι μου τι γίνεται με την προσαρμογή των αμέσων πληρωμών. να περιμένουμε στο 2019. <clears throat> και να ελπίσουμε ότι τότε θα φτάσουμε το 80%, το 85% του μέσου όρου της Ευρώπης, αυτό δεν είναι ικανοποιητικό για τους εκλογείς μας. Δεν είναι ο λόγος αυτός για τους οποίους μας έχουν στείλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν είναι ένας δρόμος ο οποίος μπορεί να είναι κατανοητός για αυτούς. Εξακολουθούν να αγωνίζονται λοιπόν οι γεωργοί μας για να υπάρξει μια δίκαια λύση. Τις επόμενες μέρες θα γίνει μια μια διαδήλωση. Στην Βία Μπάλτικα θα υπάρξει αυτή η παρουσία γεωργών. Ελπίζουμε ότι το μήνυμα αυτό θα γίνει αποδεκτό και από το Συμβούλιο και εσείς προσωπικά θα σκεφτείτε καλύτερα για όλα αυτά τα θέματα, τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί στην Ευρώπη. Είναι πολλά ερωτήματα, ελπίζω θα μπορέσετε να τους δώσετε απάντηση. Ευχαριστώ κύριε Ρούμπιξ. Περνάμε τώρα στους ε, εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές. Ο Μισελ Νταντέν πρώτα και μετά η Ράτσε Γκαρσία Πέρες. Νταντέν. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την αποφασιστικότητα που επιδεικνύεται, ούτω ώστε στου πέντε μήνε που υπολείπονται για τη μελλοντική μα συνεργασία να καταλήξετε σε ένα ικανοποιητικό για όλου ενδιαφερομένου αποτέλεσμα. Το μότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ενωμένη στη διαφορετικότητά μας. Την περασμένη εβδομάδα το Κοινοβούλιο εξέφρασε την και ε, έμπρακτα ε, ότι εφαρμόζει αυτήν την αρχή με την απόφαση που έλαβε. Όλοι έχουμε απαιτήσει, δεσμεύσει ε, σε σχέση με τι εκλογέ μα, προσδοκίε που διαφέρουν. Και όπως είπε και ο Λουίς Κάπουλα Σάντος, που είναι εισηγητής για την έκθεση για τον πρώτο πυλώνα, ήταν ευρία η πλειοψηφία με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση. Κάποιοι στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να θωρεί από αυτή τη στάση του Κοινοβουλίου. Ε, λοιπόν, πρώτη φορά η άμεση δημοκρατία εφαρμόζεται στον τομέα της ε, γεωργικής πολιτικής και ακούγεται η φωνή του λαού επιτέλους ε, στα θεσμικά όργανα που ορισμένε φορές απομακρύνονται από τους πολίτες ή ξεχνούν να τους ακούσουν. Πάντως, πώς θα ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις σε ένα πλαίσιο που είναι μάλλον παρεμφερές με αυτό που ίσχυε ε, όταν καταρτίστηκε εκείνη η γεωργική πολιτική. Πριν από 50 χρόνια που ιδρύθηκε, καταρτίστηκε πρώτη φορά αυτή η πολιτική, η Ευρώπη των 6 για όλα τα τα προϊόντα εξαρτώταν από τις εισαγωγέ. Και το πρώτο της μέλημα ήταν να κατοχυρώσει την επισητιστική ασφάλεια. 4% των ε, αγαθών που καταναλώναμε παραγάγαμε τότε. Τώρα έχουμε 500 εκατομμύρια καταναλωτές ε, και θέλουμε να εξασφαλίσουμε την επιστημιστική τους ασφάλεια, αλλά το ίδιο σημαίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι γίνεται. Ο Ευρωπαίος πολίτης περιμένει από την ε, κοινή γεωρική πολιτική μια κάποια σταθερότητα στις αγορές, μια προστασία για την τροφοδοσία, τον ανεφοδιασμό δηλαδή, προστασία σε σχέση με την ποιότητα των προϊόντων, δηλαδή πέρα από μια μια ε, λειτουργούσα γεωργία, χρειαζόμαστε μια εξίσου αισίω λειτουργούσα άγριο βιομηχανία. Γι' αυτό ζητάμε αυτά που ζητάμε στις εκθέσεις μας στην Ευρώπη 2020. Μιλάμε για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης και το επικαλεστήκατε. Λοιπόν, για το πρόγραμμα τη της Ιρλανδικής Προεδρίας, αυτό που εμείς ζητάμε είναι να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει και να επιτύχουμε την ανάπτυξη και να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Είμαστε κι εμείς αποφασισμένοι μετά από συνεργασία να καταλήξουμε σε ικανοποιητικέ συμβαστικέ λύσεις. Ξέρουμε έχουμε ψηφίσει, ξέρουμε ποιες είναι οι διαπραγματευτικές γραμμές μας για, τα διάφο... για τις διάφορες εκθέσεις. Είμαστε έτοιμοι πλέον να αρχίσουμε τις συζητήσεις. Συζητήσεις, έτσι, όχι διαπραγματεύσεις, γιατί ακόμη δεν έχουμε επίσημη διαπραγματευτική εντολή. Δηλώνω κι εγώ, λοιπόν, ότι είμαι στη διάθεσή σας, γιατί έχουμε τις ίδιες προτεραιότητες για το επερχόμενο ε, εξάμεινο. Ευχαριστούμε, Μίσελ, η Ράσε Γκαρσία Περές και Μαγκίνες και στη συνέχεια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο και εγώ θέλω να επαναλάβω τις ευχαριστίες των συναδέλφων προς τον κύριο Κόβενη για την παρουσία του εδώ και για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε κάνει σε μια στιγμή που είναι κεφαλαιώδης πιστεύω για να μπορέσουμε να φέρουμε σε περάτωση όλες αυτές τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα για την μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής με όλες αυτές τις ε, παρεμβάσεις των βουλευτών καταλάβατε και εσείς τις μεγάλες προσδοκίες που τρέφει η Επιτροπή μας για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ιρλανδική Προεδρία για να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση κοινή αγροτικής πολιτικής. Είναι σημαντικό, είναι θεμελιώδες θα έλεγα, να μπορέσουμε πράγματι να δημιουργήσουμε μια συνεργασία και ένα καλό συντονισμό για τις προσπάθειες όλων μας και ξέρουμε όλοι ότι στο Συμβούλιο μπορούν να υπάρχουν πολλές δυσκολίες όταν πρέπει να συναυτούν συμφωνίες σε ορισμένα επιμέρους σημεία. Νομίζω ότι η σύμπνοια <clears throat> και η κοινή θέση της δικής μας Επιτροπής μπορεί να είναι και ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει το Συμβουλίο να προβεί και αυτό σε ορισμένες συμφωνίες. Προφανώς και εμείς έχουμε μεγάλη πολυπικιλία, πολιτικές ομάδες και σε προέλευση από διάφορες χώρες. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει μια συμφωνία. Αλλά είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια μεταρρύθμιση η οποία θα αντιμετωπίσει τις πραγματικές συνθήκες στον αγροτικό τομέα <clears throat> και λαμβάνοντα πάντα υπόψη την πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Νομίζω ότι η διαφορά μεταξύ της αρχικής πρότασης Κομισιόν και τι θέσει που βγήκε από την Επιτροπή Γεωργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι ακριβώ λαμβάνουμε υπόψη όλε τι πτυχέ τη πολυμορφία και τι ιδιαιτερότητε που υπάρχουν στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ανάγκη διαφοροποιημένη χρήση των εργαλείων είτε στο πρασίνισμα είτε στα θέματα τη εσωτερική σύγκληση. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό και κέριο θέμα για τη δική μου χώρα. Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα των εργασιών του Κοινοβουλίου ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά προ την κατεύθυνση αυτή. Λέγατε ότι περιμένετε ότι στο τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχουμε καλά νέα και ο κύριος Φαν θα μπορέσει να δώσει κάποιες σαφείς προσδοκίες για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτές οι προσδοκίες δεν πρέπει να προκύψουν μόνο από μια συμφωνία, αλλά πρέπει να προκύψουν από μια θετική συμφωνία. Μια θετική συμφωνία θα πρέπει να σημαίνει ότι μπορούμε μέσα στα πλαίσια τη κοινή αγροτική πολιτική να μην επιφερθούν περισσότερε περικοπέ από ό,τι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν, <clears throat> σε σχέση με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή για τον Προπολογισμό τη Γεωργία, δεν πρέπει να προκύψουν σημαντικέ περικοπέ. Για την κοινή οργάνωση αγορά, νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να θέσουμε σημαντικά θέματα, τα οποία να κάνουμε προτάσει οι οποίε δεν έχουν ουσιαστικό οικονομικό κόστο. Υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με υποφελέστερο τρόπο για να ενισχύσουμε την δύναμη των παραγωγών μέσα στην αλυσίδα προσθέμενη αξία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα στη, στα θέματα ανταγωνισμού να έχουμε μια ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού και ελπίσουμε ότι και το Συμβούλιο θα αποδεχτεί αυτές τις αλλαγές που έχει εισαγάγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να υπάρξει μια συνορική συμφωνία. Και τέλος ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα, αν μου επιτρέπετε, όχι τόσο, δεν απευθύνομαι σε εσάς ως πρόεδρο του Συμβουλίου Γεωργίας, αλλά ως Υπουργό Γεωργίας της Ιρλανδίας. Πριν από δύο, δύο εβδομάδες περίπου υπήρξε μια είδηση σε σχέση με ορισμένα χάμπουργκερ που ερχόντουσαν από την ε, Ισπανία και περιείχανε κρέας αλόου. Και δεν ξέρω αν είναι σαφές σε όλους ότι αναγνώρισαν και οι ίδιες οι Ιρλανδικές αρχές ότι δεν προχώρησαν από την Ισπανία αυτά τα χάμπουργκερ, αυτό το κρέας για χάμπουργκερ. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν είναι λοιπόν σαφές ότι το πρόβλημα αυτό δεν οφείλεται στην, στην Ισπανία και κατηγορήθηκε λαθασμένα η χώρα μας για το θέμα αυτό. Αυτό είναι θέμα λοιπόν αξιοπιστίας και καλής πίστης για όλους τους παραγωγούς ε, προϊόντων αγροτικών, όχι μόνο της Ισπανίας αλλά όλη, όλης της Ευρώπης. Γι' αυτό σας ζητώ συγγνώμη γιατί είναι συγκεκριμένο αυτό το θέμα, αλλά με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, <clears throat> Ράσε. Και τώρα η κυρία Μακ και η κυρία Κώστιγκερ. Μαρία, που είσαι σκιώδης εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Με αυτό το τελευταίο σχόλιο της συναδέλφου θα κάνω εγώ μια παρατήρηση και να κάνω και ένα σχόλιο όπως και ο κύριος Νταντάν ότι θέλουμε μια διατροφική αλυσίδα που να λειτουργεί και για τους παραγωγούς και για τους ε, καταναλωτές όχι μόνο από τιμών αλλά και ποιότητας ε, σωστή σήμανση σε καταλήλων ελέγχων σε όλη την αλυσίδα ανεφοδιασμού ε, του κλάδου. Νομίζω ότι αυτές είναι οι βασικές αρχές που υπερασπίζεται η Επιτροπή μα και πρέπει να μεριμνήσουμε τους ώστε να εφαρμοστούν όλα αυτά και σε κάποια άλλη συνεδρία μπορούμε να μπούμε σε περισσότερε λεπτομέρειε. Σας καλωσορίζω και πάλι στην Επιτροπή Γεωργίας και εύχομαι να έχετε και την ίδια ενέργεια που δείχνετε σήμερα του επόμενου ε, μήνε, ε, το ίδιο και εμεί. Είναι μακροσκελέστατη η διαδικασία, αλλά δεν είναι και πυρηνική φυσική. Α σταματήσουμε, εν πάση περιπτώσει, να υπερτιμούμε περί τίνο πρόκειται. Δηλαδή, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να συμφωνήσουμε για κάποιες βασικές αρχές. Ε, όταν μιλήσατε για την επιστημιστική ασφάλεια και την περίπλοκη πρόκληση, πώς να παράξουμε δηλαδή τρόφιμα με βιώσιμο τρόπο και να αυξήσουμε και την παραγωγή μας. Σας ρωτώ λοιπόν, αυτές οι μεταρρυθμίσεις κατά τη γνώμη σας θα μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση ή όπως ε, πιστεύουν κάποιοι γίνεται μια προσπάθεια τώρα να έχουμε μια, ένα ολιστικό ε, σύστημα παραγωγής που θα ενσωματώνει και περιβαλλοντικές ανησυχίες. Ε, για να μην τα περιπλέκω, πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει αυτή η νέα προσπάθεια. Το Κοινοβούλιο έχει επιδείξει ιδιαίτερη διαλεκτικότητα μέχρι στιγμής. Έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά με τους συναδέλφους παρότι έχουμε ιδεολογικές διαφορές και μας έχετε βοηθήσει για να προχωρήσουμε και καλό είναι να συνεχίσουμε με τις άτυπες αυτές επαφές και στη συνέχεια και όταν θα αποκτήσουμε και διαπραγματευτική εντολή. Είναι καλή, καλή πίστη και λειτουργεί το Κοινοβούλιο και καλά κάνετε και μα προειδοποίησατε για το χρονοδιάγραμμα. Θα πρέπει να το σκεφτούν σοβαρά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπή, σε μια κρίσιμη φάση και θα κλείσω με το αρχικό μου σχόλιο. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Γνωρίζουμε ε, τι, ποια είναι τα εκρεμίζει και ε, ε, ε ακαθόδη ζητήματα. Πέρασε ο χρόνο ε, τη συζήτηση. Τώρα α δράσουμε και α καταλήξουμε σε μία λύση. Σα ευχαριστούμε, Ελίσσα Μπεθκιώστινγκ, τώρα που είναι σκιώδη ε, ε, εισηγήτρια για του φιλελεύθερου και θα συνεχίσουμε συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ σας καλωσορίζω κύριε Υπουργέ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ θετικά και ενθαρρυντικά σας λόγια και για τις ακριβείς απαντήσεις που δώσατε στον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Ε, και εγώ πιστεύω, και αυτό το επιβεβαίωσαν και οι προραλήσαντες ότι πράγματι είναι ένα πολύ καλό δείγμα της Ιρλανδικής Προεδρίας ότι επιθυμεί αυτές τις ε, φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις να τις ολοκληρώσει. Παρ' όλα αυτά, ετέθη το ερώτημα, και νομίζω αυτό το είπε ήδη η Κομισιόν, ότι οι μεταρρυθμίσεις ε, θα αρχίσουν να λαμβάνουν χώρα το 2015 επειδή πρέπει να υπάρξουν τεχνικές προσαρμογές. Και εγώ ερωτώ συγκεκριμένα ε, σε αυτόν τον τομέα ε, τι θα γίνει με, τις, ε, ε, με την ανάπτυξη της υπέτρου. Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει πρόβλημα με τις πληρωμές αν αναβληθεί η ημερομηνία καταβολής αυτών των πληρωμών και λόγω του ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προβούν σε προγραμματισμό, μετά να υπάρξει πιστοποίηση και δεν γνωρίζουμε ακριβώς ε, ποια θα είναι τα μέτρα πρασινίσματος. Ε, εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε καταθέσει πολύ συγκεκριμένες ε, και κατά την άποψή μου πολύ καλές προτάσεις κυρίως όσον αφορά στα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της υπέτρου. Αυτό που είναι σημαντικό είναι σε κάποια κράτη στο μέλλον να μην υπάρξει ε, οπισθοχώρηση. Και θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψή σας ε, επ' αυτού. Επίσης, με ενδιαφέρει πιο συγκεκριμένα το θέμα του προϋπολογισμού. Ε, στο, στις τελευταίες ε, διαπραγματεύσεις το Νοέμβρη παρακολουθήσαμε το τι διαδραματίστηκε και αναφέρθηκε ήδη σήμερα ότι οι ενδείξεις, κυρίως όσον αφορά το γεωργικό προϋπολογισμό, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. Η γεωργική ανάπτυξη ε, θεωρώ ότι θα πληγεί ιδιαίτερα από τις ε, περικοπές και αυτό θα έχει επιπτώσεις ε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Παρ' αυτά πιστεύω ότι το μέλλον βρίσκεται στην γεωργική ανάπτυξη, στην ανάπτυξη της υπαίθρου πρέπει να ληφθούν βέβαια υπόψη οι διαφορές και η ε, ανάπτυξη της υπαίθρου δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τις γεωργικές μονάδες αλλά ε, η ανάπτυξη αφορά το σύνολο της υπαίθρου και έτσι πρέπει να είναι. Έχουμε να ε, καλύψουμε πάρα πολλά στον τομέα της ε, γεωργικής ανάπτυξης, ε, στις υποδομές, στην εγκατάλειψη της υπαίθρου. Γι' αυτό λοιπόν με ενδιαφέρει κύριε Υπουργέ η άποψή σας, δηλαδή τι θα γίνει τελικά το Φεβρουάριο επί του θέματος αυτού και πώς θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Και ίσως μπορείτε και λιγάκι να μας ε, πείτε και κάποια μυστικά, να μας εκμυστηρευτείτε αν υπάρχει ε, ένα εναλλακτικό πρόγραμμα, αν τελικά το Φεβρουάριο δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός, ποια είναι η εναλλακτική λύση. Μήπως ε, τότε κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τελείως διαφορετικές εξελίξεις ο αντιπρόεδρος Βυσεκόφσκι και μετά Σμιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να απηχώντας την παρέμβαση του κυρίου Ρουμπίξ, να συμφωνήσω κι εγώ για τις δηλώσεις που έκανε σε σχέση με τις άμεσες πληρωμές και να προσθέσω ότι αυτή η απροκάλυπτη αδικία στα επίπεδα άμεσων πληρωμών ε, ανακράτος ε, μέλος πλήττει κυρίως ε, τα νέα κράτη-μέλη και όχι μόνο. Αυτή η ανισότητα ε, υπό το φως ε, του άρθρου 18 της Συνθήκης ε, σε σχέση με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέεται με το άρθρο 42 για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου στιγματίζεται η αδικία, η διακριτική μεταχείριση κάτι που δυστυχώς χαρακτηρίζει την ε, τρέχουσα κατάσταση. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να το δεχτούμε, διότι δεν πρόκειται μόνο για μια ανισόταμη, για μια αδικία. Πρόκειται για έκνομή συμπεριφορά σε σχέση με αυτά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία της Ένωσης. Σας ευχαριστούμε κύριε Προσεκόφσκι, ο κύριος Σμίτ και στη συνέχεια θα ξαναρχίσουμε άλλο γύρω. Ευχαριστώ Πάολο. Σάιμον, θα ήθελα να σας συγχαρώ προσωπικά και γενικότερα την Ελλαδική Προεδρία για το γεγονός ότι χρησιμοποίησατε την ευφυΐα και την ικανότητα των Κελτών σε ένα χώρο ο οποίος κυριαρχείται περισσότερο από άλλα φύλλα όπως είναι οι Γαλάτες. Είμαστε σε ένα κόσμο που σπαταλάμε και πετάμε τα 50% των τροφίμων. Εκεί είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και όχι μονάχα η προσπάθεια για την ασφάλεια των τροφίμων. Θέλω να θέσω τρία ή τέσσερα σημαντικά θέματα μαζί σου γιατί νομίζω ότι μπορεί να μα δώσει κάποια, κάποιες απαντήσεις. Έχουμε για, τις, για τους ε, στάβλους, για, τα, για την εκτροφή των ζώων. Έχουμε ζητήσει να υπάρξει κάποια πρόοδο σε αυτά τα θέματα, αλλά αλλά κράτη-μέλη εξακολουθούν να χρονοτριβούν και να καθυστερούν. Είχαμε την ε, ε, νομοθεσία για τις ε, οτόκες όνθες σε συστοιχεία κλοβών, αυτή την νομοθεσία η οποία θα έπρεπε να έχει οδηγήσει σε απαγόρευση ε, εμπορίας τροφίμων και από πουλερικά που προέρχονται από τέτοιου είδους μορφές εκτροφής. Επίσης, Επίσης είχαμε, είχε επιτροπή αυτή ψηφίσει να εξαιρεθούν οι άμεσες για τα προβατοειδή οι άμεσες πληρωμές στην Σκοτία και στην Ιρλανδία. Και εγώ θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σου για το θέμα αυτό. Και επίσης για το αλογίσιο κρέας στα μπιφτέκια, το ερώτημα που έθεσε και η Ισπανή συνάδελφος. Ίσως δεν το γνωρίζετε αυτό. Αυτό προήλθε από την ε, Ιρλανδική Υπηρεσία για τα πρότυπα τροφίμων που βρήκε ότι όχι μόνο στην Ιρλανδία αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο κυκλοφορούσαν τέτοια ε, μπιφτέκια με μέχρι 28% αλογίσιο κρέα. Αυτό δεν είναι κακό για την ανθρώπινη υγεία, αλλά δημιουργεί, διαβρώνει την εμπιστοσύνη στην αλυσίδα τροφίμων. Έχουν έρθει από την Ιταλία, από την Πολωνία, ποιο ξέρει από πού αλλού αυτό το αλογίσιο κρέας. Είναι ολοκληρωμένη η αλυσίδα τροφοδοσίας σε κρέας και αυτό το μόνο πράγμα που υπογραμμίζει είναι το αλογισιο κρέα. ειναι ολοκληρωμενη η αλυσιδα τροφοδοσία σε κρέα και απαραίτητο να είναι να είναι υποχρεωτική η ετικητοποίηση και η ανείχνευση των τροφίμων. Πιστεύω ότι πρέπει να δώσετε λοιπόν μια συνέχεια σε αυτά. Μπορεί να με επιβεβαιώσει ότι αυτό θα είναι μια προτεραιότητα για σένα. Και επίση πέραν όλο τον άλλο που έχει να, να κάνει για την κοινή αγροτική πολιτική, εγώ νομίζω ότι θα χρειαστείτε την τύχη που έχουν πάντα οι Ιρλανδοί για να μπορέσει να τα προωθήσει αυτά στο Συμβούλιο. E Dodds, λοιπόν τώρα και μετά Arkin. Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζουμε και πάλι στην Επιτροπή μας. Σας ευχόμαστε καλή τύχη στην δουλειά σας. Έχετε τεράστια ευθύνη, όχι μόνο για την κοινή γεωργική πολιτική, αλλά και για την κοινή αλληλευτική πολιτική. Είναι αυτά δύο πολύ σημαντικά θέματα. Και πολύ σημαντικά και πρέπει να επιτευχθεί πρόοδος ε, μέχρι τον Ιούνιο. Έχετε λοιπόν αντιμετωπίσετε πολλές ε, προκλήσεις ε, σε σχέση με αυτά τα δύο θέματα, τα οποία περιλαμβάνουν, έχουν σχέση βέβαια με τον προϋπολογισμό. Όμως το είδαμε αυτό σε δηλώσεις των μελών, έχουν σχέση και με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται κανείς τις προσδοκίες των κρατών μελών και των νέων και των παλιών, του βορρά, του νότου, της Ανατολής, της Δύσης. Υπάρχουν πολλές διαφορές στην Επιτροπή σχετικά με το τι πρέπει να είναι και τι πρέπει να επιτύχει η κοινή γεωργική πολιτική με ενδιαφέρον ακούω τις απόψεις για το πώς προτίθεστε να υπερπηδήσετε αυτά τα εμπόδια. Θα δείξω κάποια θέματα που έχουν σχέση με τη δική μου την εκλογική περιφέρεια στην Βορειοελλανδία. Πρώτον, περιφερειακή ευελιξία. Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε κοινή γεωργική πολιτική η οποία ε, θα καλύπτει 27 κράτη-μέλη, πόσο μάλλον όλες τις περιφέρειες ε, των κρατών μελών, με πολλές φορές ε, αντικρώμενες ανάγκες. Η περιφερειακή λοιπόν ευελιξία είναι πολύ σημαντική και με ενδιαφέρουν πολύ τα σχόλιά σας επ' αυτής. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει περιφερειακή ευελιξία και σε σχέση με το πρασίνισμα. Εγώ δεν είμαι οπαδός του πρασινίσματος στον πυλώνα 1, γιατί θα φέρει πολλά προβλήματα και ε, πολλοί από εμά λένε ότι τελικά θα καλέξουμε σε ολόκληρη γραφειοκρατία όσον αφορά το πρασίνισμα. Επίσης, ε, πρέπει και το πρασίνισμα να αντιμετωπίζεται σε περιφερειακή βάση. Αυτό θα περιορίσει ε, την γραφειοκρατία. Ξέρω ότι αυτό είναι σημαντικό και για τη δική σας την εκλογική περιφέρεια γενικότερα για την Ιλλανδία και τη Βόρεια Ιλλανδία. Αυτό το κίνημα για το σύστημα των καταποκοπή ποσών. Αυτό πρέπει να το διαχειριστούμε προσεκτικά με ένα λογικό ε, χρονικό πλαίσιο και περιμένω με αγωνία τη συζητήση στο Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Επίσης και τις ε, συζητήσεις για την ε, υποστήριξη που είναι απαραίτητη κυρίως για τους ε, γαλακτοπαραγωγούς. Έχουμε αντιμετωπίσει με πολλές αλλαγές αυτή την αγορά και κυρίως μετά το 2015 Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει υποστήριξη και δίχτυ ασφαλείας για τους γαλακτοπαραγωγούς εάν συνεχίσει αυτή η μεταβλητότητα. Ε, στην Αλία την προηγούμενη εβδομάδα αναφέρατε ότι θα γίνουν συζητήσεις στο Συμβούλιο για το θέμα των αρμοδιοτήτων, των θεσμών ε, για διάφορα θέματα και σε σχέση με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θέλω να ξέρω τι έγινε στις συζητήσεις γι' αυτό και αυτό είναι σημαντικό για μας, ε, να γνωρίζουμε με σαφήνεια. Αυτή την εβδομάδα ε, μίλησα με τον Επίτροπο Μπόρκ μετά τις ε, συζητήσεις για αυτούς τους χώρους, αυτούς τους τάβλους. Εγώ έρχομαι από μια χώρα που έχει συμβιβαστεί. Μας ενδιαφέρει λοιπόν ιδιαίτερα να γνωρίζουμε τι θα γίνει τελικά ε, και για το θέμα αυτό. Σας ευχόμαστε ε, καλή τύχη γιατί ξέρουμε ότι έχετε να αντιμετωπίσετε πολλά και δύσκολα καθήκοντα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε την κυρία Αρκίν Μπρούν και Γίγκια, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα κύριε Υπουργέ Κάβενη θέλω να σας καλωσορίσω και να σας ευχηθώ καλή τύχη. Όπως βλέπετε υπάρχει πολύ καλή θέληση για την Προεδρία σας. Όπως είπατε και εσείς είναι πολλά τα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι θέσατε το δάκτυλό σας επί των τύπων των ύλων όταν είπατε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα η Επιτροπή μας έχει προσπαθήσει να συμβάλλει σε όλα αυτά και αν δεν υπάρξει λύση σε αυτό το παράθυρο ευκαιρία, θα είναι η επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου και η επόμενη Κομισιόν που θα κλείσουν αυτές τις διαπραγματεύσεις. Κανείς δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, πρέπει να το πετύχουμε και να σταματήσουμε απλώς να μιλάμε χωρίς δράση. Επίση το θέμα τη συναπόφαση. Εμεί δεν περιμένουμε από εσά να δώσετε απαντήσει. Είναι συναπόφαση να λαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μα κι εμεί. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι τέσσερα τα θέματα που θέλω να αναφέρω. Αναφερθήκατε σε 30 εκρεμή ζητήματα. Αντί να σας ζητήσω συγκεκριμένα για τα 30 αυτά θέματα, μπορείτε να μου εξηγήσετε με τι δομές προβλέπετε να αντιμετωπίσετε αυτά τα 30 θέματα. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές προοπτικές, ακούσαμε ότι υπάρχουν προτάσεις του Φαν Ρομπάου και άλλων για σημαντικές περικοπές στις αγροτικές δαπάνες. Πώς βλέπετε αυτό να έχει αντίκτυπο στην αγροτική ανάπτυξη. Ε, μετά είπατε ότι υπάρχει ένας σε ό,τι αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Πόση ευελιξία θα θέλατε να υπάρχει για να υπάρξει διαμόρφωση του τελικού πακέτου. Και σε σχέση με τις προτάσεις που έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε δύο προτάσεις. Μία ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι 30% του εθνικού ποσού πληρωμών για να δώσει συμπληρωματικές Πληρωμέ προ του γεωργού. Αυτή είναι η γαλλική πρόταση να υπάρχει διπλή ε, πληρωμή στου γεωργού για κάποιε περιοχέ που θα καθορίσουν τα κράτη-μέλη και ήθελα να ξέρω την απόψή σα, και επίση για το θέμα του πρασινίσματο. Το Κοινοβουλίο όμω επίση δέχτηκε μια τροπολογία επί τη βάση τη οποίας το πρασίνισμα θα την χάνει μια πληρωμή που θα αποτελεί ένα ποσοστό της βασικής πληρωμής. Οπότε Κάποιοι γεωργοί θα παίρνουν διαφορετικέ πληρωμέ για το ίδιο επίπεδο πρασινίσματο. Συμφωνείτε με αυτό, ποια είναι η άποψή σα. Ευχαριστώ κύριο Λεμπρού και μετά η. Η κυρία Γέκλε. Ευχαριστώ πολύ, λέει, κυρία Λεμπρού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε δεν ε, θα ήθελα να επαναλάβω τι ευχαριστίε ε, και τι αυροφροσύνε των συναδέλφων. Συμφωνώ φυσικά και θα ήθελα όλου ιδιαίτερω να σα ευχαριστήσω για την ε, ειλικρίνειά σα. Έχουμε συνηθίσει την κυρία Μαγκίνε που ήταν εξίσου ειλικρινή κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων. Ξέρουμε ότι το επίπεδο τη συναπόφαση δεν είναι το ίδιο για όλου, παρότι ακολουθούμε μάλλον τη σωστή κατεύθυνση. Και σε αυτό εγγύεται ακριβώ και το πρόβλημα, διότι όπω είπαν και οι συνάδελφοι, και συμφωνούμε όλοι για τα διακυβεύματα τη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική, το είπατε και εσεί, η μέγιστη πρόκληση είναι η επιστημιστική ασφάλεια αλλά και η συνδιαλλαγή, η συμφιλίωση μάλλον ανάμεσα στο οικονομικό και το περιβαλλοντικό διακύβευμα. Και ε, δεν είναι σε αντίθεση αυτές οι δύο ε, συνιστώσεις, αρκεί να βρούμε την μέση οδό ούτως ώστε αντίθετα με αυτά που βλέπουμε επί να ε, συνεργάζονται αυτέ οι δύο συνιστώσει, οικονομική και περιβαλλοντική, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να τελεσφορήσει το σύστημά μας. Και το ουσιαστικότατο ζήτημα είναι τα κονδύλια και το χρονοδιάγραμμα. Όπως είπε και η συνάδελφος, και εγώ αυτή την ερώτηση ήθελα να σας κάνω, Πώς ακριβώς αποτιμάτε το επίπεδο διαλλακτικότητας ε, το οποίο θα εξευρεθεί για να καταλήξουμε συμφωνή για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δηλαδή δεν μπορούμε να υπερασπιζόμαστε τη γεωργία αλλά όχι την ανάπτυξη της υπαίθρου. Δεν έχει νόημα. Ο Μισελ Νταντά μας μίλησε για τη διαφορετικότητα στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ και εγώ, αλλά θα πρέπει να ε, εκφραστεί αυτό εμπράκτο επιτόπου. Αυτό περιμένουν από εμά οι γεωργοί η, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά είναι όντως διαφορετικά, αλλά θα πρέπει να ισχύσουν και διαφορετικοί κανόνες ε, για τις διάφορες εκμεταλλεύσεις ε, και να προστατευτούν οι μικρές εκμεταλλεύσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Η Ελίζαμπεθ και στη συνέχεια Γκίρλινγκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω και για αυτά τα οποία είπατε μας δώσατε την εντύπωση ότι έχετε σαφείς στόχους που θέλετε να πετύχετε με έναν τρόπο ο οποίος είναι συνεκτικός και συστηματικός. Εάν εμείς θέλουμε να έχουμε σταθερότητα επί τη βάση της αηφορίας και θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη, επί αυτής της βάσης αυτό είναι ένας εφικτός στόχος. Εγώ θα ήθελα όμως να σταθώ εδώ περισσότερο στο δεύτερο πυλώνα της αγροτικής πολιτικής εσείς κατανοείτε από αυτά που είπαμε ότι και οι δύο πυλώνες είναι σημαντικοί. Ο πρώτος για τη γεωργία αυτή καθεαυτή, αλλά ο δεύτερος αφορά τη συνολική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και την σωστή κατεύθυνση των δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό που αφορούν και άτομα πέραν των γεωργών. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο έχει κάποιες δυσκολίες στις τωρινές συζητήσεις. Όπως είπε ο πρόεδρός μας ότι αν μας επικρίνουν όλες οι παρατάξεις και όλες οι πλευρές, τότε οι προτάσεις μας δεν μπορούν να είναι και τόσο άσχημες. Χθες ήμουν στη Νότια Γερμανία και συνάντησα γεωργούς και εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι είχαν μια θετική άποψη για τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν λοιπόν μπορεί να μειωθεί η γραφειοκρατία και αν μπορούν να εφαρμοστούν ε, ικανοποιητικά αυτές οι ρυθμίσεις νομίζω ότι θα είναι αποδεκτές και στους γεωργούς. Το δικό μου <coughs> πρόβλημα είναι ότι ζητήθηκε όχι μονάχα να αντιμετωπίζονται οι οικολογικές εκμεταλλεύσεις ως ε, πράσινες, αλλά και αυτές οι οποίες εδώ και πολλά χρόνια ακολουθούν οικολογικά μέτρα και να τύχουν και αυτές μια ισοδίκαιας μεταχείρισης. Αυτό ήταν και η δική μας θέση στην ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' αυτό καταλήξαμε στη λύση της διπλής χρηματοδότησης σε ορισμένες περιπτώσεις. Ορισμένοι βλέπουν κάτι το αρνητικό στην διατύπωση διπλή χρηματοδότηση, αλλά αυτό σημαίνει απλώς ότι θέλουμε ορισμένες μορφές επιχειρήσεων να την χάνουν τη ισοδίκαια μεταχείρισης όπως και οι οικολογικές εκμεταλλεύσεις. Δεν είναι λοιπόν επομένως μια διπλή χρηματοδότηση, επομένως μια ευνοϊκή μεταχείριση για ορισμένους, αλλά μια διόρθωση για να εξασφαλίσει την ίση μεταχείριση για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος, Ελίζαμπετ. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτά που έχουμε κάνει. Γκίλιν και μετά ο αντιπρόεδρος κύριος Σεκεριέσκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να χαιρετήσω την παρουσία του κύριου Κόβεν. Είναι πολύ σημαντικό που είναι εδώ παρόν μαζί μας. Δεν θα μιλήσω για την κοινή αγροτική πολιτική, ίσως αυτό σας ανακουφίσει λιγάκι. Νομίζω ότι τα ίδια πράγματα λέγονται και επαναλαμβάνονται. Θα περάσω τώρα σε κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι υπάρχει εδώ ένα κίνδυνο ότι μπορεί να λησμονήσουμε άλλα σημαντικά θέματα. Θα ήθελα να σταθώ σε μια ανακοίνωση της Κομισιόν από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών στις 20 Ιανουαρίου που περιείχε μια πρόταση για κάποιες μορφές παρασιτοκτόνων που έχουν να κάνουν με το μελισσοκομικό τομέα. Πολλοί από αυτά που εργαζόμαστε στον τομέα αυτών ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα σε ερευνητικό επίπεδο για αυτά τα παρασιτοκτόνα και απαντήσεις οι οποίες θα πρέπει να δοθούν για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα να ξέρω αν η Γενική Διεύθυνση υγειονομικών και καταναλωτικών θεμάτων ακολουθεί μια αναλογική μεταχείριση στα θέματα αυτά. Για να σας υπενθυμίσω, υπάρχει μια πρόταση από 1η ε, Ιουλίου να υπάρξει απαγόρευση νεονικοτινοειδών παρασιτοκτόνων, αλλά συγχρόνως αναγνωρίζεται ότι δεν υπάρχουν σαφείς επιστημονικές εμπειρογνωμοσύνες, ότι η πραγματομοσύνη αυτή έγινε βεβαιασμένα και επίσης ότι είναι πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των ε, ε μελισσών, όπως είναι οι μονοκαλλιέργειες, όπως είναι άλλοι ε, βιολογικοί παράγοντες. Επομένως, το ερώτημα είναι ότι δεν είναι αναλογικό για μένα να υπάρξει μια απαγόρευση αυτών των νέων οικοτινοειδών παραστοκτώνων, γιατί επίσης ένα μέρος του προβλήματος προέρχεται από την κατάχρηση αυτών των ε, ουσιών. Φαίνεται ότι αυτοί οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα παραστοκτόνα με σωστό τρόπο έχουν δει ωφέλη από τη χρήση τους. Υπάρχει αύριο μια συνάντηση, σήμερα, συγγνώμη, σήμερα, για τα θέματα αυτά και η απόφαση θα ληφθεί με Εξτελεστικέ πράξεις. Μόνο το Συμβούλιο επομένως θα αποφασίσει για τα θέματα αυτά. Το Κοινοβούλιο δεν εμπλέκεται. Εγώ θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι δικές σας για το θέμα αυτό, εάν μπορείτε. Και πώς νομίζετε ότι θα προχωρήσει αυτή η συζήτηση με τη Σκόφα και κατά πόσο το Συμβούλιο έχει κάποια άποψη για τα θέματα αυτά. Νέο και Ευχαριστώ. Για τα παρασιτοκτόνα, τα οποία αναφερθήκατε κι εσείς, ε, το σημαντικότερο ζήτημα είναι το εξής. Εάν καταργήσουμε τα παρασιτοκτόνα, ποια είναι η αναλλακτική μας λύση και σε ποιο βαθμό θα μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το χειρότερο είναι να δεν έχουμε τα απαιτούμενα δεδομένα στη διάθεσή μας. Υπολείπεται σοβαρό το έργο για να ολοκληρώσουμε τις γνώσεις μας. σα επανέλθω τώρα στην μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πρασίνισμα, παρεμβάσεις, ε, αυτές είναι οι κύριες γραμμές της μεταρρύθμισης. Δηλαδή παρεμβαίνουμε άμεσα στην παραγωγή και στα εισοδήματα των παραγωγών. Εάν λοιπόν επιθυμούμε την παρέμβαση θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ταυτόχρονα και κάποιο αντιστάθμισμα για αυτή την παρέμβαση. Πρόκειται για ένα κονδύλι που για την επόμενη περίοδο θα μειωθεί κατά 12%. Ε, οι βαλτικές χώρες έχουν χαμηλότερο επίπεδο άμεσων πληρωμών. Θα έπρεπε λοιπόν να απορροφήσουμε κονδύλια από αυτούς που λαμβάνουν υψηλά ποσοστά βοήθειας για να τα επαναδιοχετεύσουμε στις ε, νέες χώρες που λαμβάνουν χαμηλότερη βοήθεια. Αυτό φυσικά δεν θα μπορέσει να προβλεφθεί ποτέ στους όρους προσχώρησης ε, σε περίπτωση νέων κρατών μελών. Η μεταρρύθμιση θα εκλειφθεί από τους ε, γεωργούς ως συρρήκνωση των κονδυλίων. Δηλαδή θα έχουν στα χέρια τους λιγότερα χρήματα η παραγωγή επίθεση ε, κατά του δευτέρου πυλώνα θα χτυπήσει ε, την Ήπεθρο όπου υπάρχει και η μεγαλύτερη ανάγκη για επενδύσεις ε, στην υποδομή και τα γεωργικά μηχανήματα. Επεξεργαζόμαστε λοιπόν τον κανονισμό για το 2014, όμως δεν είμαι καθόλου σίγουρος εάν θα καταφέρουμε ε, στο τέλος ε, να επιτύχουμε μια ικανοποιητική μεταρρύθμιση. Φοβούμαι ότι θα είναι πολύ χαμηλή σε ποιότητα, αν κρίνω από τα αποτελέσματα μέχρι τούδε. Θα είναι, όπως ε, είπα και στην αρχή της παρέμβασής μου, μια μεταρρύθμιση παρεμβατική. Αυτή η παρέμβαση είναι και η άμεση απόρρια των φυσικών διακυμάνσεων που εκφεύγουν και του ελέγχου των γεωργών. Δηλαδή η συγκομιδή μπορεί να αυξομοιωθεί κατά 10-15% για λόγους που ε, εκφεύγουν του ελέγχου των γεωργών. Η παρέμβαση λοιπόν είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λήθους ε, της κοινή γεωργικής πολιτικής όσον αφορά στην αγορά. Για την ε, πολιτική συνοχή τώρα, Έχουμε την εντύπωση ότι ακολουθείται η ίδια κατεύθυνση όπως και με την πολιτική της ανάπτυξη υπαίθρου και υπάρχουν ε, ε, τμήματα της υπαίθρου που είναι πραγματική ουραγή. Νομίζω ότι από στρατηγικής πλευράς ε, πρόκειται για ένα σοβαρότατο σφάλμα διότι ήδη βλέπουμε τις ε, αρνητικές επιπτώσεις αυτής της πολιτικής και πάντοτε τίθεται το ζήτημα των εξωτερικών ε, σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μας ακούει ο υπόλοιπος κόσμος όταν ε, μιλάμε για το μέλλον της επιστημιστικής ασφάλειας, αλλά ίσως να τα αφήσουμε αυτό το ε, σημείο για κάποιο μελλοντική συνεδρίαση. Αλλά δεν μπορούμε να απουσιάζουμε. Πρέπει να αγωνιστούμε και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Αλλά δεν αρκεί ε, ό,τι κάνουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε, Αντιπρόεδρε. Ας ακούσουμε την κυρία Σάντρα Καλνιέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα όπως και άλλοι συνάδελφοι να επιβεβαιώσω ότι ε, έχουμε μεγάλες προσδοκίες για την Ιρλανδική Προεδρία αλλά αυτό προϋποθέτει ότι θα έχουμε συμφωνία για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και για την κοινή γεωργική πολιτική. Εάν δεν πληρούνται αυτές οι δύο προϋποθέσεις, τότε η συμφωνία θα αναβληθεί μέχρι την επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Καλή επιτυχία πάντως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δράζεται επί κάποιων βασικών αρχών, μεταξύ των οποίων είναι η ενιαία αγορά και ο δίκαιος ανταγωνισμός στο εσωτερικό αυτής της αγοράς. Κάθε φορά που συζητώ με γεωργούς στη Λετωνία και στις άλλες δύο βαλτικές χώρες με ρωτούν πάντοτε για ποιον δίκαιο ανταγωνισμό μιλάς και για δεν ισχύει για μας. Ο Πρωθυπουργό μα. στο Συμβούλιο έχει αυτή την κόκκινη γραμμή. Χρειαζόμαστε μία δίκαιη λύση και για τον πρώτο και για το δεύτερο πυλώνα ε, για τη Λετωνία αλλά και για τη Λιθουανία και την Εστονία θα έλεγα ότι υπάρχει η ίδια αποφασιστικότητα να καταλήξουμε σε συμφωνία. Καταλαβαίνω επίσης ότι τα χρήματα που χρειαζόμαστε για την ε, συνοχή θα αφαιρεθούν ε, από τις επιδοτήσεις προς άλλες χώρες. Όμως, η γεωργοί των άλλων αυτών χωρών, μην ξεχνάτε ότι εδώ και δεκαετίες είχαν την ε, οικονομική ευκαιρία να οικοδομήσουν μια, ένα ισχυρό γεωργικό τομέα. Οι τρεις βαλτικές χώρες όμως όχι. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης καταφέραμε, ε, κατάφεραν μάλλον να φτιάξουμε μια ελεύθερη κοινή οργάνωση αγοράς ε, με όλες τις επιπτώσεις ε, που γνωρίζουμε. Ελπίζω να καθοδηγήσει τις διαπραγματεύσεις με τρόπο ώστε να είναι δίκαιη η τελική λύση. Ευχαριστούμε οι δύο τελευταίες παρεμβάσεις, και Χίγκινς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε προς ενημέρωσή σας. Ε, θέλω λιγάκι να ε, αμβλύνω τις ε, προσδοκίες της Επιτροπής σε σχέση με τον προπλογισμό. Και μιλώ με την ιδιότητά μου του μέλους του προπλογισμού. Είναι αλήθεια ότι ο κύριος Βαν ελπίζει να επιτευχθεί συμφωνία στις 7 και 8 Φεβρουαρίου. Θέλω όμως να σας υπογραμμίσω ότι αν τελικά ή αν θέλουμε να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία, ακόμα υπολείπονται πάρα πολλά. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ακόμα και αν το Συμβούλιο στις 7 και 8 Φεβρουαρίου επιτύχει συμφωνία, με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας, η συμφωνία αυτή πρέπει να εγκριθεί από το σύνολο των Ευρωβουλευτών. Και το συντομότερο που μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο είναι στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Εκεί πρέπει να υπάρξει ειδική πληροφορία πλειοψηφία. Οι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι το Κοινοβούλιο ε, έχει πολύ υψηλές ε, προσδοκίες ε, όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. 550 υπερψήφισαν 1,13 αύξηση. Αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου και θέλω να σας υπενθυμίσω αυτό απέχει πάρα πολύ από την πρόταση του κυρίου Βαν Χομπέη. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο έχει ορίσει τέσσερα βασικά σημεία, τέσσερα βασικά αιτήματα και τα τέσσερα αυτά αιτήματα δεν είναι αποδεκτά αυτή τη στιγμή από το Συμβούλιο. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι κατά πάσα πιθανότητα το Κοινοβούλιο τελικά να, θα, να απορρίψει την πρόταση του κυρίου Βαν Χομπέη το Μάρτιο. Και αν αυτό συμβεί, τότε θα έχουμε κατά το μέγιστον τρεις μήνες για να καταλήξουμε σε συμβασμό. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ε, δεν υπάρχουν καθόλου ενδείξεις για το τι τελικά θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα για την κοινή γεωργική πολιτική. Πολύ ωραία, Ρίτσαρτ, πολύ καλά έκανες ε, και μας τα υπενθύμισε όλα αυτά ο κύριος Ντόρφμαν που δεν ήταν στον κατάλογο, ε, τελευταίος ομιλητής και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό. Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε ο συναδελφός μου, δηλαδή στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν πρόκειται μόνο για τα χρήματα, γιατί με τα χρήματα συνδέονται και συγκεκριμένα θέματα. Και αν δει λίγο τις ε, προτάσεις, δεν πρόκειται για το συνολικό ποσό το ο προϋπολογισμός ε, αποτελείται από γραμμές οι οποίες και αυτές ε, έχουν ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Γι' αυτό λοιπόν σαφώς και μπορεί να συμβεί με την απόφαση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο σημαντικά τμήματα της γεωργικής μεταρρύθμισης ε, να αποφασιστούν de facto από τους Υπουργούς Γεωργίας και εμεί απλά να τους κυνηγάμε από πίσω. Γι' αυτό λοιπόν Θέλω να μου πείτε, εσείς πώς πιστεύετε ότι συνδέονται αυτά τα δύο. Όσον αφορά τώρα το περιεχόμενο της γεωργικής μεταρρύθμισης, πολύ σωστά είπατε ότι στόχος μας πρέπει να είναι μια μεταρρύθμιση η οποία ε, κατά την ε, επόμενη δεκαετία θα είναι ανταγωνιστική στην Ευρώπη και ε, θα είναι προσανατολισμένη και στο μέλλον. Αν το επιθυμούμε αυτό, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε ε, με κουράγιο. Αυτή τη στιγμή περίπου το 80% του συνόλου των δαπανών στην κοινή γεωργική πολιτική προέρχονται από χρήματα φορολογουμένων που χρησιμοποιούνται για να στηριχθεί το εισόδημα των γεωργών και το 20% των κονδυλίων χρησιμοποιούνται κυρίως στον δεύτερο πυλώνα για να καταστεί η γεωργία ε, καινοτόμα να προαχθούν οι επενδύσεις και ούτω καθεξής. Όμως ε, πρέπει να σας πω ότι δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε από αυτά τα ποσά. Ε, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πώς η γεωργία πραγματικά στο μέλλον μπορεί να είναι περισσότερο καινοτόμα. Και το είπαν αυτό αρκετοί συνάδελφοι σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία αντιμετωπίζουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή, οβιδιακή αλλαγή. Κατά την, ε, η δεν, είναι πλέον, ε, δεν έχει αγορά ε, προσφοράς αλλά ζήτησης. Και αυτό αποτελεί μια ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με την πολιτική που εφαρμόσαμε μέχρι σήμερα, όπου το θέμα ήταν τι θα κάναμε με αυτό το πλεόνασμα των τροφίμων στην ευρωπαϊκή αγορά. Και εδώ απευθύνομαι κυρίως στη δική σας την προσωπική θέση ως Υπουργού της δικής σας της χώρας. Πάρα πολλοί προλαλήσαντες είπαν ότι στο θέμα της εσωτερικής της σύγκλησης θα έπρεπε να προχωρήσουμε με μεγαλύτερο θάρρος. Ε, υπάρχει μια προσπάθεια ε, από κρατημέλη που στηρίζουμε, δηλαδή ε, να προχωρήσει αυτή η ιστορική σύγκληση και να σώσουμε όσα μπορούν να σωθούν. Αλλά αυτή η προσέγγιση δεν είναι προσανατολισμένη στο μέλλον. Στη Γερμανία αλλά και γενικότερα στις γερμανόφωνες περιοχές υπήρχε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η έννοια, ο όρος του γεωργού του σαλονιού. Δηλαδή γεωργοί οι οποίοι είχαν ε, αγροκτήματα, τα εκμίστοναν και ζούσαν πάρα πολύ καλά. Καθόντουσαν στο σαλόνι τους, ε, στον καναπέ τους, ε, άλλοι παρήγαγαν το γάλα και αυτοί είχαν απλά το όφελος. Αν δείτε λοιπόν την κατάσταση σε ορισμένες χώρες και αυτό αφορά και τη Γερμανία. Ξέρετε τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή τίνουμε στο να δημιουργήσουμε μια κατηγορία γεωργών πάλι σαλονιού που ζουν με τις επιδοτήσεις. Οι γεωργοί λοιπόν οι οποίοι έχουν αυτές τις ε, επιδοτήσεις, όμως κατ' ουσίαν έχουν απομακρυνθεί από τη Γεωργία και με αυτές τις επιδοτήσεις ζουν πάρα πολύ καλά. Αυτό λοιπόν το γνωρίζει η κοινή γνώμη, έχει προκαλέσει κριτική και θεωρώ ότι όλα αυτά θα μπορέσουμε να τα ελέγξουμε μόνο εφόσον απομακρυνθούμε το συντομότερο δυνατόν από αυτές τις ιστορικές, αυτές τις επιδοτήσεις και περάσουμε σε ένα άλλο μοντέλο το οποίο θα είναι περισσότερο γενικευμένο και θα αφορά περισσότερους. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Higgins. Πριν όμως το πράξω αυτό, να καλωσορίσω μία ομάδα Ιρλανδών φοιτητών που ήταν εδώ σήμερα το πρωί και είναι μέλη της ε, Ένωσης Young Fin Girls δηλαδή ε, είναι πρόσκυντες στον Υπουργό μας και γι' αυτό τους χαιρετώ εδώ και δίνω το λόγο στον τελευταίο μιλητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Μαγκίνες ε, τους προσκάλεσε και τους έφερε εδώ πέρα. Είναι η πολιτική του μέλλοντος ε, αυτή η νέη, όπως και οι υπόλοιποι ομιλητές. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό Κόβενη. Ε, ήσασταν Ευρωβουλευτή για τρία χρόνια. Καλωσορίσατε και πάλι στο Κοινοβούλιο. Ε, λοιπόν, ε, για την κοινή γεωργική πολιτική και την κοινή αλληλευτική πολιτική έχετε ευθύνη ταυτόχρονα, οπότε χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας έχουμε εδώ. Ε, σας θαυμάζω, είσαστε πάρα πολύ φιλόδοξο στους στόχους και στο χρονοδιάγραμμα που θέσατε για την Ιρλανδική Προεδρία και με ευελπιστούμε ότι θα συμβούν όλα όπως θα έχετε προβλέψει. Τρία σημεία εν συντομία. Πρώτον, για τον πυλώνα 1 και τον πυλώνα 2. Ε, πιστεύετε ότι θα υπάρξει ευελιξία σε σχέση με αυτούς τους δύο πυλώνες. Δεύτερο ζήτημα, η αποσύνδεση. Ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη που δεν έχουν αποσυνδέσει τις επιδοτήσεις τους ε, δεν θα είναι σε ε, δυσμενέστερη θέση. Και τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, περιφερειοποίηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Εγώ πιστεύω δεν θα έπρεπε ε, να χρησιμοποιηθεί αυτό και να καταργηθούν τα ιστορικά σημεία αναφοράς για τον υπολογισμό των πληρωμών. Και να ευχαριστήσω κλείνοντας και πάλι την κυρία Μαγκίνας. Ωραία, τελειώσαμε αυτή την μακρά σειρά παρεμβάσεων. Αγαπητέ Σίμων, και τώρα έχει δυνατότητα να απαντήσεις και σε ευχαριστούμε εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας. Καλή εργασία, έχουμε πολλές κοινέ ευθύνε. σε αυτή την ελλαδική Προεδρία και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε καλό αποτέλεσμα. Έχεις το λόγο για να κλείσεις. Ε, ε, πολλές ερωτήσεις κρύβονταν πίσω από τα τελευταία σας λόγια και δεν θέλω να σπαταλίσω το χρόνο σας. Θα προσπαθήσω όμως με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στις διάφορες απαντήσεις που θα σας δώσω. Μπορώ να εκφράσω την προσωπική μου άποψη με την ιδιότητα του Ιρλανδού Υπουργού, αλλά μην ξεχνάτε ότι εδώ έχω διπλό καπέλο όπως λέμε, δηλαδή με προεδρεύω και στο Συμβούλιο ε, οπότε εκφράζω και τις απόψεις του Συμβουλίου. Είναι σημαντικό λοιπόν εξ αρχής να κάνουμε αυτόν τον ε, διαχωρισμό. Τα πρώτα σχόλια που έγιναν από τον κύριο Ρούμπιξ και άλλους εξάλλου συναδέλφους ε, που, από βαλτικές χώρες. Λοιπόν, θα έλεγα τα εξή. Πήγα στη Λετωνία, Λιθουανία και Εσθονία και έμεινα στο καιρό πριν από λίγου μήνε στο Βίλνιου, στη Ρίγα και στο Τάλιν. Θέλω πραγματικά να προσπαθήσω να καταλάβω το γεωργικό σύστημα, γιατί ήξερα εξ αρχής ότι θα ήταν ζήτημα αυτό και είναι. Από Ιρλανδικής Σκοπιάς υποστηρίζουμε ε, τις εκκλήσεις των τριών χωρών ε, για μεγαλύτερη σύγκληση ως προς το επίπεδο ε, άμεσων πληρωμών. Αρχικά θα δούμε αυτό το ζήτημα στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και στη συνέχεια θα το διαπραγματευτούμε με το Κοινοβούλιο. Κανείς δεν πρέπει να θεωρεί οτιδήποτε δεδομένο Πιστεύω ειλικρινά ότι για αυτές τις τρεις χώρες η τελική τους θέση θα είναι καλύτερη από την αρχική βάση της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, δεν θέλω όμως να δώσω συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Ε, γνωρίζετε όλοι πόσο, ε, ποια είναι η επικρατούσα τάση, δηλαδή ε, με, με τα κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή όλοι αναγνωρίζουν την ανάγκη ότι πρέπει να υπάρξει μια εξίσωση, αλλά δεν θέλω να έχουμε υπερβολικές προσδοκίες και τελικά την επόμενη εβδομάδα να ε, μην απαλληθευτούν αυτά από τους αρχηγούς ε, κρατών και κυβερνήσεων. Ε, πάντως κατανοούμε και συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας. Όμως χρειάζεται και ένα αντιστάθμιμα. Μιλάνε όλοι για την ισότιμη μεταχείριση. Ωραία, πρέπει όμως να εξορροπήσουμε και τους δύο πυλώνες, διότι είναι διαφορετικές οι πρικοδοτήσεις για τους δύο πυλώνες, ανά ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης Τη υπαίθρου και σε αυτές τις χώρες ε, και θα πρέπει λοιπόν να το δείτε σφαιρικά, δηλαδή η σύστημα στήριξη κοινή γεωργικής πολιτική για τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, αλλά σε ε, αυτό είναι ένα συνδυασμό τη λειτουργία ε, των δύο πυλώνων, όπω σα έλεγα. Ε, κάποιες ε, χώρες θα έχουν αυξήσει στον πρώτο πυλώνα και αυτό θα πληρωθεί από άλλες χώρες που χάνουν κατά μέσο όρο. Είναι ένα ε, πρότυπο προσέγγισης. Ε, έχετε το 90% των πληρωμών και όλοι φτάνουν τα δύο τρίτα της μέσης βοήθειας, αλλά δεν γίνεται αυτό να υλοποιηθεί αν δεν αφαιρεθούν κονδύλια από κάποιους. Σε αυτό το πρότυπο βασίστηκε, σε αυτό το μοντέλο υπολογισμού βασίστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποθέτω ότι αυτό είναι το πρόβλημα με τις βαλτικές χώρες, διότι υπολείπονται πολύ του μέσου όρου άμεσων πληρωμών. Ε, γνωρίζετε την προσωπική μου άποψη, όμως οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα λάβουν την τελική πολιτική απόφαση και το Κοινοβούλιο θα κληθεί στη συνέχεια το Μάρτιο να εγκρίνει ή να απορρίψει αυτή τη θέση των αρχηγών. Μισελ έκανε μια κατά σημαντική δήλωση, δηλαδή είμαστε ενωμένοι στην επικοινομορφία. Μα ναι, είναι κοινή στρατηγική των 27 και σύντομα 28 κρατών μελών της Ένωσης, όμως θα πρέπει να γίνει σεβαστό το ότι ανάμεσα στην Κύπρο και τη Βόρειο Φινλανδία έχουμε πολλές και διαφορετικές καλλιεργητικές μεθόδους, αγροβιομηχανίες ε, και προκλήσεις ως προς την ανάπτυξη της υπαίθρου. Είτε μιλάμε για την ε, άρδευση, για τα δάση, για τους Λεόνες, ε, ε, ισχύουν διαφορετικά δεδομένα και θα πρέπει Όντω να έχουμε μια κοινή πολιτική, όμω προσοχή. Δεν πρέπει να απομακρυνθούμε τόσο πολύ από την κοινή πολιτική και να γίνουμε τόσο ευέλικτο ώστε να, κάνει, να πράττει κατά το δοκούν κάθε κράτο, ε, διότι έτσι χάνουμε την κοινή προσέγγιση σε σχέση με την παραγωγή τροφίμων, που κατά τη γνώμη μου θα οδηγήσει σε εντελώ το ανταγωνισμό στην ε, κοινή αγορά. αγορά. Δηλαδή είναι μια άσκηση ισορροπία. Να διατηρήσουμε την ενιαία αγορά και την κοινή πολιτική και να έχουμε κοινά πρότυπα για την παραγωγή τροφίμων ταυτόχρονα θα σεβόμαστε την ποικιλομορφία και την ανάγκη για ευελιξία, ούτω ώστε να λειτουργήσει ένα τέτοιο κοινό σύστημα. Το Κοινοβούλιο έχει καταβάλει σημαντικέ προσπάθειε για να επιτύχει ακριβώ αυτή την ισορροπία μέσα από τι συμβαστικέ λύσει που πρότεινε. Δεν ήταν εύκολο. Θα ήθελα τώρα να σχολιάσω ε, το θέμα του αλογίσιου αλόγου στα χάμπουργκερ. Ένα ε, ένα σκάνδαλο που ξέσπασε πριν από δύο εβδομάδες είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε. Ε, στην Ιρλανδία ε, εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν θα εκτιλοδεικτούσε κανείς στην Ισπανία και καταλαβαίνω πόσο ευαίσθητοι είσαστε γιατί πέρσι είχαμε και το θέμα με τα αγκουράκια και καταλογίστηκε αυτό στην Ισπανία με εντελώ άδικο και αναλυθή τρόπο. Ε, τι συνέβη λοιπόν. Έχουμε την ε, αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων που εξαρτάται από το Υπουργείο Γεωργίας, ε, το δικό μου Υπουργείο δηλαδή στην Ιρλανδία και κάνουν δείγματοληπτικούς ελέγχους στα καταστήματα που πουλούν τα χάμπουργκερ ως μέτρο δηλαδή προστασίας των καταναλωτών. Εδώ και καιρό κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Και πήραν τα αποτελέσματα από ένα φτηνό κατεψυγμένο ε, το φθηνότερο κατεψυγμένο κρέας για χάμπουργκερ ε, και ήταν ε, κάποια συστατικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του κρέατος και εντοπίστηκε και αυτό το ποσοστό του κρέατος που προέρχεται από τα άλογα. Ε, τα ολοκληρωμένα αποτελέσματα ελέγχου έδειξαν ότι τα συστατικά στοιχεία που βρήκαμε σε άλλες ε, χώρες ε, που έχουν στοιχεία DNA υποειδών βρέθηκαν και στην Ιρλανδία. Δηλαδή δόθηκαν διάφορες εξηγήσεις σε σχέση με το αν προέρχεται το κρέα από αυτέ τι χώρε, ή συνέβη κάτι στη μεταφορά. Πάντως για λόγους διαφάνειας έκριναν ότι έπρεπε να δημοσιεύσουν ε, όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων και σε αυτό το πλαίσιο, στο ανακοινωθέν τύπο, αφέρθηκε η Ισπανία και μία άλλη χώρα. Μεταγενέστεροι έλεγχοι δε κατέδειξαν με σαφήνεια ότι η ουσιαστική πηγή του προβλήματο ε, που ήταν ένα πολύ σημαντικό ε, τμήμα DNA υποειδών ε, προερχόταν από ένα άλλο κράτος μέρος. Και στο Υπουργείο μου ποτέ δεν δακτυλοδεικτούσαμε την Ισπανία, ποτέ δεν το κάναμε αυτό. Ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί και περιμέναμε να έχουμε καταλητικά στοιχεία. Τώρα τα έχουμε, παρεμπιπτόντως. Ε, εάν λοιπόν υπήρξε οποιαδήποτε σύγχυση ή ε, πέρασε μια αρνητική εικόνα στην Ισπανία, λυπούμε, δεν ήταν ουδόλως η πρόθεσή μας. Ήθελα να ξεκαθαρίσω, πάντως η Ισπανία δεν ήταν η πηγή του προβλήματος, ούτε και η Ολλανδία, που ήταν ε, το άλλο κράτος που αναφέρθηκε στο αρχικό ανακοινωθέν τύπου. Ε, Όμω υπήρχε λόγος που έγινε αυτή η μία για λόγους διαφάνειας Σα είπα για να δημοσιευθούν όλα τα αποτελέσματα ελέγχου και έχουμε τα ίχνοστοιχεία από ε, το, τους ελέγχους που κάνουμε για το DNA και εντοπίζονται τα πάντα στα πάντα, γνωρίζετε, με, αυτά, με αυτούς τους ελέγχους και χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος τώρα για τα συστατικά των τροφίμων ε, και έτσι ε, αναφέρθηκε ως πιθανή πηγή αυτή η χώρα. Ζητώ συγγνώμη αν δημιουργήθηκαν δυσκολίες στη χώρα σας. Λυπούμεθα πολύ, δεν ήταν καθόλου η πρόθεσή μας. Με κοίταξε σαν το φιλιτάκι για τη Μαρία Μαγκίνες. Είπατε ότι είναι ποινική φυσική αυτά πάντα Δεν είναι. Ούτε αστροφυσική. Είναι μια διαπραγμάτευση. Έχει να κάνει με την ε, περάτωση μιας συζήτησης, μιας διαπραγμάτευσης η οποία γίνεται για πολλά χρόνια. Δύο χρόνια με τρόπο έντονο και προπαρασκευαστικά δύο χρόνια. Θα δοκιμαστεί λοιπόν η διαπραγματευτική ικανότητα του επόμενου πέντε μήνε και ελπίζουμε θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια πραγματιστική λύση για να μπορέσουμε να φέρουμε το πλοίο αυτό ει ασφαλή λιμένα. Πιστεύω λοιπόν ότι με τον τρόπο αυτό θα δείξουμε κάποια θετικά αποτελέσματα γιατί συλλογικά θα είναι μια μεγάλη καταστροφή να μην τελειώσει αυτή η εργασία μέχρι το τέλος του Κοινοβουλίου. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά δεν είναι αστρονομία αλλά αλλά δείχνουν ότι θέλουμε πράγματι να προχωρήσουμε και να πραγματοποιήσουμε όλους αυτούς τους στόχους, ιδίως αν φτάσουμε στους τριγωνικούς διαλόγους, γιατί αυτό νομίζω ότι θα μας αναγκάσει μέσα σε 10 εβδομάδες να κάνουμε κάτι το οποίο κανονικά χρειάζεται 18 μήνες στη φυσιολογική διαδικασία. Αυτό δεν είναι απλό. Για την ασφάλεια των τροφίμων, αν θα λειτουργήσουν όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι μπορούν να λειτουργήσουν αλλά έχετε και εσεί την ίδια ευθύνη που έχουμε και εμεί και εγώ για να εξασφαλιστεί αυτό επί τη βάση των τροπολογιών που έχετε διατυπώσει και των θέσεων που έχετε αναλάβει όλοι από, από κοινού θα πρέπει να επιτύχουμε τη σωστή εξισορρόπηση μεταξύ τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων που τηρεί τι επιστημονικέ ε, ε, βάσει και συγχρόνω να εξασφαλίσουμε την ανάκαμψη όπω είναι απαραίτητο για να έχουμε την απαραίτητη τροφιμική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνάτε ότι εξακολουθούμε να εισάγουμε πάρα πολλά τρόφιμα στις χώρες μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να διαφρέψουμε τον πληθυσμό μας. Για την Ελίζαμπεθ αναφερθήκατε στις μεταβατικές ρυθμίσεις. Νομίζω ότι κάποιο από την Κομισιόν θα σα παρουσιάσει τα θέματα αυτά με πολύ περισσότερα λεπτομέρεια. Εμεί δεν έχουμε δει ακόμα την πρόταση τη Κομισιόν σχετικά, αλλά ο αρμόδιο επίτροπο προτίθεται να κάνει μια πρόταση για το πώς θα μπορέσουμε στο 2014 να έχουμε μεταβατική εφαρμογή κανονισμών και ρυθμίσεων που θα ισχύσουν από το 2015. Όλα αυτά είναι πραγματιστικά μέτρα. Και αυτό είναι όμω ο λόγο για τον οποίο εμεί πρέπει να εστιάσουμε στο να πάρουμε τώρα τι απαραίτητε πολιτικέ αποφάσει, ώστε να έχουμε χρόνο να κάνουμε όλα αυτά που είναι απαραίτητα υπομορφή μεταβατικών μέτρων για το 2014 και όλων των άλλων συναφών μέτρων για το κοιτίο διαπραγματεύσεων στις ε, πολιετής ε, δημοσιονομικές προοπτικές. Ναι, είναι αλήθεια αυτά τα οποία λέγονται για την ε, αγροτική πολιτική. Εγώ μπορώ να πω εξ ονόματο του Συμβουλίου ότι θέλουμε ένα ισχυρό προπολογισμό για τα γεωργικά θέματα για τα επόμενα 7 χρόνια. Ξέρετε όμως ότι αυτό είναι ότι είναι κομμάτι της γενικής διαπραγματεύσης μεταξύ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που προσπαθούν να εξισορροπήσουν τον προπολογισμό τη στιγμή που πολλοί ισχυρέ χώρε επιμένουν να περικοπεί ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ προσωπικά συμφωνώ απόλυτα με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά αναγνωρίζω και τι πραγματικότητε, τι πολιτικέ που αντιμετωπίζουν πάρα πολλέ χώρε σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό του. Και αυτό είναι το γενικό πλαίσιο το οποίο θα λειτουργήσει για μια συμφωνία για τι πολιτικές δημοσιονομικέ προοπτικέ. Κύριε Αντιπρόεδρε, νομίζω ότι πολύ σωστά είπατε για τι βαλτικέ χώρε ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι δεν νιώθουν να είναι θύματα διακρίσεως αυτές οι χώρες μετά την διαδικασία αυτή. <clears throat> Και ο Άλεν μας έδωσε και κάποια ανακούφιση για ορισμένα θέματα για την ε, στέγαση των χειρομητέρων ο Επίτροπος Μπότς είχε κάνει σαφές ότι η Κομισιόν τώρα θα προχωρήσει προς την εφαρμογή των κανόνων εναντίον κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται. Όλοι καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει τώρα να συμμορφωθούμε το ταχύτερο δυνατό. Βέβαια, δεν έφτασε να πει ο κύριος Επίτροπος ότι θα πρέπει να υπάρξει απαγόρευση εμπορίας προϊόντων από παραγωγούς που δεν έχουν εφαρμόσει όλες τις προδιαγραφές. Φαντάζομαι ότι αυτό που θα λάβει η χώρα είναι ότι η Κομισιόν θα προχωρήσει προς την εφαρμογή των κανόνων αυτών με τις χώρες που εμπλέκονται και αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία γρήγορα και τα 6 ή 7 κρατημέλη που δεν έχουν φτάσει ακόμα σε 100% συμμόρφωση θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό πάρα πολύ προσεκτικά μετά από τις προθέσεις αυτές που ανέφερε η Κομισιόν. Για το σύστημα εντόπισης και ανείχνευσης των ζώων έχουμε μια συμπεφωνημένη θέση του Συμβουλίου για όλα αυτά, αν το Κοινοβούλιο αλλάξει τη θέση του για τα θέματα αυτά, τότε θα πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων δεν μπορώ τώρα να σας δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση για το θέμα αυτό. Προσπαθώ να είμαι επακριβής σε αυτά που λέω. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει αποφασίσει το Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά. Για την ε, σήμανση προέλευσης και την ε, διαμάχη σε σχέση με το αλογίσιο κρέας, έχουμε μια δέσμευση από την Κομισιόν να εισαγάγει αυτή τη σήμανση προέλευσης για το κρέας με έναν τρόπο που είναι συμβατός με αυτά τα οποία ισχύουν ήδη για το βόλιο κρέας και για το, τα πουλερικά, για το αρνίσιο και χείριο κρέας Όλα αυτά είναι μια κίνηση προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά ξέρει το Κοινοβούλιο ότι έχουμε να κάνουμε πολλά περισσότερα ακόμα και πρέπει να προχωρήσουμε για τα θέματα αυτά. Εγώ εξ ονόματος του Συμβουλίου δεν μπορώ να δεσμευτώ αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρω πόσες είναι οι ανησυχίε που δημιουργήθηκαν με αυτή την υπόθεση πάλι. Η Νταϊάν μίλησε για την διαχείριση των προσδοκιών στα κρατη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό για εμά ω Υπουργού στο Συμβούλιο αλλά και για εσά ω Ευρωβουλευτέ να διαχειριστείτε σωστά τις προσδοκίες των γεωργών στις χώρες μας. Ας μιλήσουμε λησμονούμε ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του εισοδήματος των ε, γεωργών που βασίζεται στην ε, κοινή αγροτική πολιτική και τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα. Πολλοί γεωργοί δεν θα μπορούσαν να παραμείνουν ενεργοί χωρίς την κοινή αγροτική πολιτική. Επομένως, πράγματι, στα αγροκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει πολλή ανησυχία για τα θέματα αυτά και εγώ προσπάθησα να διοργανώσω δημόσιες συζητήσεις όπου να εξηγήσω τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τα πιθανά αποκοίηματα αυτής της διαδικασίας για τους γεωργούς. Και όπως είπε και ο Γερμανός ή Αυστριακός συνάδελφός μου, είναι λογικη η γεωργη είναι άνθρωποι που καταλαβαίνουν άμα τους εξηγήσει κανείς τι γίνεται ή τι δεν γίνεται. Αυτό που δεν θέλουν είναι να τους δημιουργείτε διαγκωμένες προσδοκίες και στη συνέχεια να μην μπορείτε να τις στηρίσετε αυτές τις υποσχέσεις. Σε ό,τι αφορά την ευκαμψία μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα, θα υπάρξει κάποια ευελιξία. Ξέρω ποιε είναι οι απόψει σα. Εμεί προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια συνολική θέση του Συμβουλίου για τα θέματα αυτά. Χρειάζεται να υπάρχει κάποια ευελιξία και χρειάζεται να υπάρξουν και πολλέ συζητήσει για τα θέματα των ισοδυνάμεων. Η πρόταση της Κομισιόν αυτή τη στιγμή είναι ότι αν είσαστε βιολογικός γεωργός, αυτόματα παίρνετε την πληρωμή για το πρασίνισμα. Πολλές χώρες θα ήθελαν να υπάρχουν και άλλες κατηγορίες γεωργών που θα είναι αυτοδικαίως ε, συστήματα πρασινίσματος, είτε είναι για το πρακτικές περιβάλλοντος ή κάτι άλλο. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε σύντομα να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα σε τα θέματα αυτά στο Συμβούλιο. Αναφερθήκατε και την υποστήριξη για τη γαλακτοκομική παραγωγής. υπάρχουν θέματα τα οποία θα ανακύψουν μετά το 2015. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να κάνουμε προφανώ. Προσωπικά όμω, ξέρετε ότι οι γεωργοί ξέρουν ότι θα σταματήσουν οι γαλακτοκομικές ποσοστώσει. το ξέρουν εδώ και πολύ καιρό και γι' αυτό δεν θα πρέπει να, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να έχουμε ένα συστηματικό τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούμε το τέλος των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Τα διαθεσμικά θέματα. Αυτό ενδιαφέρει και την ΚΑΠ, αλλά ενδιαφέρει και την αλληλευτική πολιτική, την κοινή αλληλευτική πολιτική. Τη Δευτέρα συζητήσαμε για πρώτη φορά στο Συμβούλιο για τα θέματα αυτά και εγώ χαίρομαι που υπήρξε μια θετική προσέγγιση, αλλά όπως και στο Κοινοβούλιο υπάρχουν στεναρές απόψεις, υπάρχει και στο Συμβούλιο μια στεναρή απόψη για το τι σημαίνει η συνθήκη Λισαβόνας για τα διάφορα θεσμικά όργανα. Εγώ δεν ζήτησα να υπάρξει μια εντολή από τους ομολόγους μου. Απλώς ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψη των κυβερνήσεων και των υπουργών για το τι μπορούν και θέλουν να συζητήσουν και να και τώρα στην Προεδρία να φέρει προτάσεις στον τομέα αυτό για το πώς μπορούμε να προωθήσουμε το θέμα αυτό με ένα τέτοιο τρόπο ώστε η κοινή αλληλευτική πολιτική και η κοινή γεωργική πολιτική να προχωρήσουν. Αυτό το θέμα χρονίζει εδώ και δύο χρόνια και υπάρχουν θέσεις οι οποίες είναι αμετακίνητες. Αλλά ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουμε και θα βρούμε κάποια λύση από αυτές τις θέσεις οι οποίες είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εδρεωμένες. Ενίσχυσε το μήνυμα ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρία ε, η κυρία Χάρκιν σε σχέση με τα τρία εκκρεμή ζητήματα. Με ρωτήσατε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, η δική μου δουλειά είναι να τα ρυθμίσω αυτά τα ζητήματα πρώτα απ' όλα στο Συμβούλιο. Και είναι πολύ δύσκολο αυτό ε, για μένα πραγματικά. Ε, θα εστιάσω την προσοχή μου σε αυτό. Ταυτόχρονα θα έχουμε και άτυπε συζητήσει για να προετοιμάσουμε του τριμερεί διαλόγου. Για να πετύχετε κάτι πρέπει να έχετε ένα σχέδιο για να το πετύχετε, έτσι. Και αν συμβεί κάτι καθοδόν που σα υποχρεώνει να αλλάξετε το αρχικό σα σχέδιο, ε, τι να κάνουμε τώρα. Ε, αυτό έγινε και με, τις, ε, με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εάν το Μάρτιο θα δούμε ότι δεν γίνεται, ε, θα ε, επανασταθμίσουμε τη θέση μας, θα αλλάξουμε το αρχικό μας σχέδιο και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περάσει το ζήτημα σε μελλοντική προεδρία, ε, τι να κάνουμε και πάλι. Αλλά πρέπει να, κάνουμε, να βασιστούμε σε κάποιες υποθέσεις για να μπορέσουμε να καταρτήσουμε ένα σχέδιο και για να πετύχουμε κάτι. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει το Μάρτιο για την ψηφορία τη δικιά σας στην Ολομέλη θα δούμε τι θα γίνει στο Συμβούλιο. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε τίποτα, αλλά πρέπει να υποθέσουμε ότι αν τελικά εγκριθεί αυτό από το Κοινοβούλιο, θα προλάβουμε να καταλήξουμε σε τελική απόφαση τον Ιούνιο. Αν όλα τα κάνετε βήμα-βήμα και δεν βασίζεστε σε κάποια δεδομένα, δεν προχωράμε και δεν θα υπάρχει ποτέ αρκετό χρόνο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ε, και γι' αυτό αρχίζουμε από, την, από το αποτέλεσμα. Δηλαδή λέμε τι θα θέλαμε εν τέλει, μία πολιτική απόφαση επί της αρχής ή και στην πράξη τον Ιούνιο και το παίρνουμε αντίστροφα. Δηλαδή για να φτάσουμε και τον Ιούνιο τι πρέπει να γίνει από, στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Έτσι φτιάξαμε τον οδικό χάρτη για την ε, Προεδρία μας για να επιτύχουμε αυτά που θέλουμε να επιτύχουμε. Σε σχέση με το συγκεκριμένο σας ερώτημα για το, ε, για το ευέλικτο πρασίνισμα. Εάν ε, υπάρχει διαφοροποίηση των πληρωμών ανά εκτάριο στους ε, γεωργούς ε, στην ίδια χώρα είτε σε επίπεδο περιφερειοποίησης είτε σε εθνικό επίπεδο τότε θα πρέπει να βασίζεται στην ίδια, στο ίδιο κριτήριο για το πρασίνισμα. Είναι απλό να πούμε ότι το 30% όλων των πληρωμών θα είναι πρασίνισμα. Όχι να πούμε το 30% του μέσου όρου πληρωμών της χώρας αυτής θα αντιστοιχεί στο πρασίνισμα. Είναι στο μίξ της συζήτησης για το πρασίνισμα. Δεν έχει αποφασιστεί αυτό ακόμα για την ε, ε, γαλλική πρόταση για τα πρώτα 15 εκτάρια η καταποκοπή, οι επιπρόσθετες πληρωμές, ε, ούτε αυτό έχει ολοκληρωθεί. κυρία Λεμπρά, με ρωτήσατε. στη χρηματοδότηση ανάπτυξη υπαίθρου θα υπάρξει ευελιξία. ελπίζω ναι, σε σχέση με το παρελθόν. Πιστεύω ότι πολλοί υπουργοί, κυβερνήσεις και βουλευτές ε, νιώθουν απογοητευμένοι σε σχέση με το πώς ε, λειτουργούσε μέχρι στιγμής το σύστημα του δεύτερου πυλώνα για τις στρατηγικές δαπάνες. Λοιπόν, ε, η νέα προσέγγιση για, την, για τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων, δηλαδή για την βιωσιμότητα, για την βιοπικιλία, Ελπίζουμε ότι θα δώσει μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων στις κυβερνήσεις και γενικότερα στους πολιτικούς, ε, ούτως ώστε να αποκομίσουν μεγαλύτερα ωφέλεια από την πολιτική ανάπτυξη υπαίθρου, ακόμη και τα μέτρα πρασινίσματος ε, και η σχέση ανάμεσα στους δύο πυλώνες ε, είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να εξετάσουμε ως ιονή πηγή ευελιξίας. Οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες παραδείγματος χάρη είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ την Επιτροπή σας, η υποστήριξη προς τους μικρούς καλλιεργητές το ίδιο. Η Ελίζαμπεθ μας μίλησε για την βιολογική γεωργία, για τον ορισμό του πρασινίσμου κτλ. Νομίζω ήδη έδωσα κάποιες τμηματικές απαντήσεις για αυτά τα ζητήματα. τώρα, ως προς το... Ένα λεπτάκι. Α, ναι. Τα επικριτικά σχόλια ε, που έρχονται από όλες τις πλευρές. Μα καλό σημάδι είναι αυτό, σημαίνει ότι ε, ακολουθούμε μια ε, ισόρροπη προσέγγιση. Για την επόμενη ερώτηση, δηλαδή σε σχέση με την απάντηση του ΣΚΑΦΚΑ από πλευρά Επιτροπή και Συμβουλίου. Σήμερα συνεδριάζουν και πήρα ένα feedback από αυτέ τι σκέψει. Χρειαζόμαστε ισορροπία ανάμεσα στην ανάληψη δράσης βάσει επιστημονικών δεδομένων αφενός και αφετέρου μια προληπτικής προσέγγισης ε, για τα νοικοτινοειδή δεν νομίζω να ισχύσει πλήρη απαγόρευση. Τμηματική ίσω για κάποιε καλλιέργειε που τραβάνε όλο ιδιαίτερο τι μέλισσε. Αυτό ναι αλλά συνολική απαγόρευση όχι. Θα βρούμε λοιπόν μια ε, ισορροπία, θα γίνει και ψηφοφορία. Στο Σκάφκα θα περάσει μετά το θέμα στην ε, Κορεπέρ. Το συζητήσαμε ε, την περασμένη Δευτέρα στην Κορεπέρ και επιζητείται ισορροπία από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξαναλέω, να δρούμε επί τη βάση της αρχή τη πρόληψη, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να απαγορεύσουμε κάποια νοικοτινοειδή, νέο νοικοτινοειδή, ε, διότι δεν έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας όλα τα επιστημονικά δεδομένα. Θα περιμένουμε λοιπόν να γίνει έλεγχος και θα δούμε. Ε, σε σχέση με τις βαλτικές χώρες νομίζω έχω ήδη απαντήσει. Στον επόμενο γύρο των συνομιλιών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου θα πρέπει να εξεταστεί και αυτό το ζήτημα. Ο Ρίτσαρτ Άσουαρτ χαίρομαι που είναι εδώ, διότι μας υπενθύμησε λιτά όλες τις προκλήσεις που περιστρέφονται γύρω από τις πολιετές δημοσιονομικές προοπτικές. Για την Επιτροπή Γεωργίας και το έργο της και το συλλογικό μας έργο υπάρχει μεγάλη σύνδεση με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλά Ξέρετε, σε αυτό το διαπραγματευτικό κοιτίο υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες για την κοινή γεωργική πολιτική πέρα από το θέμα της χρηματοδότησής της. Μην το ξεχνάτε αυτό. Θα ήθελα ε, να ε, συνειδητοποιήσετε το πόσο επίγον είναι αυτό το ζήτημα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο με τρόπο πολιτικά αποδεκτό για αυτό, να εισαγάγετε όλα αυτά τα στοιχεία για την κοινή γεωργική πολιτική, ούτω ώστε να καταφέρουμε ε, να καταλήξουμε συμφωνία το Μάρτιο. Θα κλείσω, θα κλείσω, Πρόεδρε, ξέρω δεν έχουμε χρόνο. ο Χέρμπερ Ντόρφμαν μου έκανε επίση μια ερώτηση. Ξέρω ότι έχετε ιδιαίτερες ανησυχίες για την υποστήριξη των ενεργών γεωργών και τη συμμερίζομαι, αλλά τώρα να με γενικεύσουμε τη χρήση των καταποκοπή πληρωμών δεν νομίζω ότι λύνει το πρόβλημα της γεωργίας. Ε, αυτό το θέμα του γεωργού του καναπέ, ε, του σαλονιού, ε, δεν έχει σχέση με την, ε, το επίπεδο της ε, πληρωμής, έχει σχέση με το είδος της πληρωμής και κάποιοι ισχυρίζονταν ότι οι άμεσες πληρωμές συνδέονται με τους μεγάλους γεωργούς που έχουν μεγαλύτερη επιλεξιμότητα, είναι ενεργοί γεωργοί, έχουν μεγαλύτερες καλλιέργειες. Η, το, η συζήτηση της εσωτερικής σύγκλησης είναι ένα ζήτημα καυτό ε, κάποιες χώρες που έχουν επιλέξει τις καταποκοπήν πληρωμές θέλουν ε, να ακολουθήσουν και όλες οι υπόλοιπες χώρες. Οι υπόλοιπες χώρες δεν θέλουν. Ε, χρειάζεται μια συμβαστική λύση. Χρειάζεται συζήτηση και σε εσάς και σε εμάς για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Καλωσορίζω τους προσκεκλημένους του Φίνα Γκέιλ χαίρομαι που σας βλέπω εδώ πέρα. Α, ο Τζέμις ε, με ρώτησε για την ευελιξία ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο πυλώνα. Θα υπάρξει ευελιξία γιατί θα υπάρξει και αποσύνδεση και επαναλαμβάνω ότι ε, όσες χώρες έχουν διατηρήσει σε δεδομένες πληρωμές ε, θα έχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες για την σύνδεση. Όσες έχουν αποσυνδέσει τελείως πληρωμές τους και θέλουν να, να γενικεύσουν την αποσύνδεση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να κάνουν και εκείνες κάποιες υποχωρήσεις, να βρούμε και πάλι τη μέση οδό. Για την περιφερειοποίηση είναι σημαντικό για τα τελικά βασικά αποτελέσματα των συζητήσεών μας να εξασφαλίσουμε ότι θα δώσουμε εναλλακτικέ λύσεις, δηλαδή θα επιτρέψουμε στις χώρες, στις διάφορες περιοχές στις χώρες να εφαρμόζουν πιο ειδικέ λύσεις, όπως παραδείγματος χάρη και στην Ιρλανδία ισχύει και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, είναι πολύ διαφορετικές ε, οι ανάγκες ανάλογα με το είδος των καλλιδιών και των εκμεταλλεύσεων και άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα περίπλοκα προβλήματα ε, προσφέροντας εναλλακτικέ λύσεις. Το συγγνώμη, αλλά ήταν πάρα πολλά τα ερωτήματα ερωτήματα και κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ειλικρίνειά σας ε, ή ακόμη και την ομότητά σας θα έλεγα και ευχαριστώ και τον πρόεδρο για τον τρόπο με τον οποίο κατήφθηνε τη συζήτηση ε, και ε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό ο τρόπο που χειριστεί κατά θέμα τη κοινή γεωργική πολιτική του τελευταίου μήνε και ελπίζω να βγούμε αληθινοί παρά τι υψηλέ προσδοκίε μα και να συνεχίσει η καταπληκτική αυτή συνεργασία. Ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ε, πολύ καλά ξεκίνησε η Ιρλανδική Προεδρία. Τώρα λοιπόν, συνάδελφοι, πρέπει να περάσουμε στο σημείο υπαριθμών 5. Είναι η παρουσίαση εκ μέρου τη Επιτροπή ε, των Μεταβατικών Διατάξεων για τι μεταρρυθμίσει στο πλαίσιο τη ΠΑΚ. Έχουμε μιλήσει με την Επιτροπή, με τον κύριο Πλέμπε κυρίω. Αυτό το επιχείρημα νομίζω ότι αφορά όλου. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διαθέση μας, γι' αυτό και προτείνω να αναβληθεί το θέμα αυτό για την επόμενη συνεδρίαση που όπως ξέρετε θα είναι στις 20-21 Φεβρουαρίου. Είναι ένα επιχείρημα, ένα θέμα το οποίο απαιτεί να υπάρξουν ερωταπαντήσεις. Ας το αναβάλουμε λοιπόν αυτό το θέμα για την επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και για άλλη μια φορά ε, την Ιρλανδική Προεδρία. Λύει τη συνεδρίαση.